Good afternoon. Καλησπέρα σας. Ας συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σημεία της μερίσιας διάταξης. Για σήμερα το απόγευμα, ως κεντρικό θέμα, έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Χάν. Προφανώς τον καλωσορίζουμε για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Προπολογισμών, από τότε που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως Επίτροπος για θέματα προπολογισμού από την 1η Δεκεμβρίου του 2019. Καταλαβαίνετε ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας και για την Επιτροπή βέβαια την Ευρωπαϊκή, γιατί βρίσκεται υπό εξέταση και διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα αποτελέσει την ακρογωνία λίθο για τις στρατηγικές προκλήσεις που έχει προτείνει η πρόεδρος Φοντρε Στην ακρόασή σα τον Οκτώβριο, κύριε Χάν, είπατε ξεκάθαρα ότι οτιδήποτε βρίσκεται ή υπολείπεται μάλλον των προτάσεων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτεύστημα αστυνομικό πλαίσιο θα είναι ζημιογόνο για την ε, φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποδυναμώσει την ικανότητα της Ένωσης να καταλήξει σε απτά αποτελέσματα. Είπατε επίση ότι ε, ήταν εφικτό να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων. Προσβλέπουμε λοιπόν στην παρέμβασή σας να δούμε τι έχετε να μας πείτε για τα ζητήματα αυτά, καθώς επίσης και για άλλα ζητήματα. Τώρα, στο ενδιάμεσο διάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να μας αποκαλύπτει σιγά-σιγά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα μας παρουσίασε το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και το επενδυτικό σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία. Τώρα, η χρηματοδότηση του μηχανισμού αυτού και η διασύνδεσή του με το τρέχον πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλου ιδιαίτερα στα μέλη τη Επιτροπή μα. Μία από τι αποστολέ σα επίση φέτο θα είναι να επιβλέψετε την εφαρμογή του τελευταίου προπολογισμού του τρέχοντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και να προτείνετε ένα νέο προσχέδιο προπολογισμού για το 2021. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα είναι όλο και πιο επίγον να έχουμε ένα σχεδιασμό έκτακτη ανάγκη στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε εγκαίρω να συμφωνήσουμε για το πολιτέ νομοσυνομικό πλαίσιο. Δυστυχώ, βέβαια, εξαιτία τη καθυστέρηση που έχει σωρεύσει τα τελευταία δύο χρόνια το Συμβούλιο. Προτού δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χάν για να κάνει την εισαγωγική του παρέμβαση, να του ζητήσω να περιοριστεί στα 10 λεπτά και εν συνεχεία αυτό που σας προτείνω να πάρουν το λόγο οι συντονιστές και όχι οι πρέσβεις όπω είπε ο Πρόεδρος, ενδεχομένως κάποια μέρα <laughs> να γίνουν και πρέσβεις, κανείς δεν ξέρει πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, σας προτείνω να... διαφορετικά από ό,τι σήμερα το πρωί, να έχουμε πέντε λεπτά για κάθε παρέμβαση, να θέσετε δηλαδή την ερώτησή σας ή την παρατήρησή σας και να απαντήσει με στο πεντάλεπτο ο Επίτροπος. Αφού ακούσουμε τους συντονιστές, θα δοθεί προφανώς και δυνατότητα και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας να πάρουν το λόγο, με προτεραιότητα βέβαια στους συζητητές για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον προπολογισμό του 2021. Στην περίπτωση βέβαια αυτή θα πρέπει να αφιερώσουμε τρία λεπτά στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Του το λεχθέντον έχετε το λόγο κύριε Χάν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου υπενθυμίσατε ότι επισήμωση είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας. Βέβαια δεν το είχα αντιληφθεί γιατί σας συναντώ τόσο συχνά που δεν μου είχε περάσει καν από το μυαλό. Πάντως ε, και εγώ εύχομαι να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δεν θα εξαντλήσω το δεκάλεπτο γιατί νομίζω ότι συζητούμε συνεχώς αυτά τα θέματα ε, και δεν ε, θα ήθελα να ε, μην αναφερθώ κι εγώ σε αυτά τα οποία εσείς είπατε και ο προκατοχός μου, ο κύριος Έτιγκερ και η συνολική προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσπαθούσαμε να προωθήσουμε την πολιτική στοχοθέτηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πάντοτε με βάση τους υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σίγουρα έχουμε τις επιπτώσεις για το Brexit και σίγουρα η απόφαση, μάλλον η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί επιτάπητος δεν έχει πέσει από τον ουρανό, δεν είναι κάτι άξαφνο. Ε, σίγουρα ε, υπάρχει επίσης και μια νέα δυναμική. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι δεσμευμένο και προσιλωμένο στη λήψη αποφάσεων ε, και για το Συμβούλιο ελπίζω επίσης να υπάρχει ειλικρίνεια ε, και ιδίω από πλευρά του Προέδρου του Συμβουλίου, του κυρίου Μισελ, να υπάρχει λοιπόν ε, η εντολή για το Συμβούλιο. Υπάρχουν επαφές με τα κράτη-μέλη και φυσικά και εγώ ως αρμόδιος επίτροπος ε, είμαι προσιλωμένος σε αυτή την προσπάθεια. Θα μεταβώ και εγώ στις διάφορες πρωτεύουσες, στα κράτη-μέλη για να καταθέσουμε σε μια ξεκάθαρη θέση και θα δω και τι διαφορετικές απόψεις υπάρχουν και πρέπει να σας πω ότι σύντομα πάω στη Στοκχόλμη, αυτή είναι η πρώτη μου επίσκεψη. Είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι και εγώ θέλω να τους πετύχουμε ε, και σίγουρα θα το πω ξεκάθαρα και στα κράτη-μέλη ότι έχουμε την ξεκάθαρη στάση και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι στην Επιτροπή Προπολογισμών είναι πολλοί βουλευτές που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία από προηγούμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και σίγουρα υπάρχει το θέμα και της ευελιξίας, ε, υπάρχει το θέμα των ιδίων πόρων και σίγουρα οι ε, πολύπυροι βουλευτές ε, που έχουν διαπραγματευτεί στο παρελθόν το προηγούμενο πιδελταπή και τους προϋπολογισμούς μπορούν να συνεισφέρουν τα μάλα στον τομέα αυτό για να σημειωθεί σημαντική πρόοδος και όποια κράτη έχουν επιφυλάξεις ε, θα πρέπει ουσιαστικά να τους πούμε ότι δεν θα πει ότι ο προϋπολογισμός ε, είναι ένα μόνο μία πηγή και θα προέρχονται τα έσοδα ε, από μία μόνο και οι δαπάνε θα καθορίζονται από μία μόνο πηγή. Ούτε αυτό σημαίνει όμως ότι ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν πάρα πολλές ε, ε, θυσίες και να μεγαλώσουν πολύ τις εισφορές τους. Το Δεκέμβριο υπήρξε από τη Φιλανδική Προεδρία ένα nego box, ένα διαπραγματευτικό κουτί, και ξέρετε ότι υπάρχουν ε, διάφορα ε, ποσά που φτάνουν μέχρι και τα δις ε, στις, στο τέλος της δεκαετίας. Έχουμε το 1,67 που... αυτά που είναι μια βελτίωση, αλλά θα πρέπει σίγουρα να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που προέκυψαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει περικοπές ουσιαστικά για να λάβει υπόψη όλες ε, τις ευστίες στον τομέα, παραδείγματος χάρη της γεωργίας, ε, στον τομέα της συνοχής ε, και να ληφθούν υπόψη και άλλοι σημαντικοί πολιτικοί τομείς όπως είναι το πράσινο σύμφωνο, η ψηφιοποίηση, η μετανάστευση και ασφάλεια έρευνα και καινοτομία και να μπορέσουν και εκεί να διατεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια. Η πρόταση της ε, Φινλανδικής ε, Προεδρίας ε, ουσιαστικά ψηλοαλλάζει πάλι κάπως τα πράγματα, αλλά με τη δική σας την υποστήριξη Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις για την ευελιξία και για το σύστημα ιδίων πόρων και μάλιστα να ε, επιμείνουμε περισσότερο σε αυτό το νέο σύστημα. Είχαμε τη μεταναστευτική κρίση, ε, δεν την αντιμετωπίσαμε ε, ή δεν την είχαμε μάλλον ε, προβλέψει και αν δεν υπήρχε ευελιξία δεν θα την αντιμετωπίσαμε με τον τρόπο με τον οποίο καταφέραμε να την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει και ένα σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω. Ίσως δεν έχει συζητηθεί πολύ, αλλά αν δούμε τις διάφορες κατηγορίες, τους διάφορους τίτλους, ε, τα διάφορα heading και το διοικητικό κόστος ε, μειώνεται κατά δύο δις. από 75 δις. Σε τρία μπλοκ θα μπορούσα να το ομαδοποιήσω. Μιλάμε για το διοικητικό κόστος ε, ε, των θεσμικών ε, οργάνων και των εκτελεστικών οργανισμών. συνολικά είναι το 6,7% του προϋπολογισμού και σίγουρα πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε ως το δυνατόν πιο αποδοτικοί Έχουμε τις συντάξεις κατά ένα τρίτο, το τρέχον κόστος ένα τρίτο, ενέργεια, ε, μισθώματα κτλ. Ε, και μισθή ε, το τρίτο, τρίτο αν μπορώ να το πω έτσι. Έχουμε τρία μπλοκ δηλαδή. Εμείς μόνο στους μισθούς ουσιαστικά μπορούμε να επηρεάσουμε γιατί για τις συντάξεις ε, ε, και την ενέργεια, τα ενισθώματα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς. Πρόκειται για μακροχρόνιες μισθώσεις ε, και τα λοιπά. Οπότε έχουμε ουσιαστικά το 1 τρίτο στο οποίο θα πρέπει να επιβληθεί αυτή η μείωση κατά 2 δισεκατομμύρια ε, που σημαίνει ουσιαστικά η οποιαδήποτε συνταξιοδότηση δεν θα μπορεί να οδηγεί σε αντικατάσταση του ή της απερχόμενης υπαλλήλου για τα θεσμικά όργανα και δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε έτσι να ε, προχωρήσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ ε, στοχευμένη προσέγγιση και το πώς θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα. Πάντως ε, νομίζω ότι σε αυτό το διαπραγματευτικό κουτί υπάρχουν και κάποια θετικά, πολύ θετικά, ότι παραδείγματος χάρη πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει αυτό το ποσό 25%. Ε, επίσης η προστασία του κράτους δικαίου και το σχετικό κριτήριο. είναι κάτι σημαντικό που λαμβάνεται υπόψη. Ο μηχανισμός δικής μετάβασης, ε, εδώ πιστεύω ότι συζητήσατε εντατικά την προηγούμενη εβδομάδα, εβδομάδα ε, η πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε μία πρώτη αναφορά σε ό,τι αφορά αυτή τη σημαντική χρηματοδότηση των 7,5 δισεκατομμυρίων που θα είναι νοπό χρήμα το οποίο θα έλθει να προσθεθεί στα εφιστάμενα κονδύλια για την δίκαιη μετάβαση έγινε όπως είπα πολύ συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα οπότε δεν φαντάζομαι ότι ε, χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεσμεύεται να στηρίξει πλήρως την Κροατική Προεδρία ε, και σε αυτήν την προσπάθεια και θα εμβαθύνει και τι επαφέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και ήταν εδώ ο Πρόεδρος Μισελ, μίλησε μαζί σε αυτό, είναι θεωρώ πολύ θετικό και ο Κροάτης Επαρχουργός κ. Πλένκοβιτ επίσης τοποθετήθηκε. Οπότε τώρα νομίζω ότι έχουν τεθεί, έχει τεθεί το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και Θα πρέπει τώρα να ε, καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική για όλους ε, λύση. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτό το οποίο ανέφερε και ο Πρόεδρος, ε, τον λεγόμενο προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης, το contingency planning. Εγώ θέλω να σας επαναλάβω κάτι. Νομίζω ότι Αυτό που είναι βασικός μας στόχος είναι το πι και η τελευταία, η έσχατη περίπτωση είναι να ε, έχουμε αυτό τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης. Ε, νομίζω ότι αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε από εδώ και πέρα είναι να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε ε, για να τελειώνουμε με το ΠΔΠ. Εκεί θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Και δεν νομίζω ότι ήδη από τώρα είναι ανάγκη να αρχίσουμε να εξετάζουμε έναν μηχανισμό εκτακτής ανάγκης. Πάντως πρέπει να σας πω ότι ε, εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα ε, να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Και ε, το είδατε και εγώ τέλο πάντων κάπω στο περιθώριο ίσω, αλλά είδα πόσο καλά λειτουργήσε η συνεργασία μα και για την κατάρτιση του προπολογισμού του 2020. Ε, όσοι με γνωρίζουν θα ξέρουν ότι η πόρτα μου είναι πάντοτε ανοιχτή. Οπότε πραγματικά θα υπάρχει δυνατότητα για διμερείς επαφές ε, και συνομιλίες μεταξύ μας, ωστόσο, ώστε να επιλύσουμε ε, τα ζητήματα της χρηματοδότησης ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις πολύ σημαντικές ε, πολιτικές και την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και εμείς και το είναι και Γενικός Διευθυντής εδώ θα είμαστε έντιμοι διαμεσολαβητές, honest brokers σε αυτή την προσπάθεια και σίγουρα υπάρχει και το θέμα του διαχείριση των προσδοκιών, expectation management. Ε, το πρόβλημα ε, δεν είναι να βρίσκουμε τι μας χωρίζει, αλλά πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τις απόψεις και να έρθουμε πιο κοντά ε, τα διάφορα θεσμικά όργανα. Και αυτός είναι ο στόχος μας και για το πολιτές μας. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Επίτροπο για την παρουσία του αλλά και για τη δέσμευσή του και για όσα είπε στην ε, ακρόαση. Είναι σαφές ότι η παλαιά θέση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, αποτελεί το ελάχιστο για τούτη την Επιτροπή. Ε, λέω, αναφέρομαι στην παλαιά θέση της Κομισιόν, γιατί με την Πράσινη Συμφωνία, καθώς και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει ε, να υπάρξει επικαιροποίηση, τουλάχιστον από τεχνικής απόψεως, έτσι ώστε να ξαναδούμε λίγο τα αριθμητικά στοιχεία. Υπάρχουν νέες εμπλοκές, νέες προτεραιότητες και οπωσδήποτε και νέες προτεραιότητες ε, οι οποίες χρήζουν πόρων, επιπλέον προσθέτων πόρων, όσον αφορά το ζήτημα των κρατών μελών που θέλουν να μειωθούν οι διοικητικές ε, ε, δαπάνες. Αυτό αποτελεί παγίδα στην οποία δεν θέλουμε να πέσουμε εμείς, είναι λαϊκισμός. Για να πούνε δήθεν στους πολίτες, ορίστε, καταβάλλονται προσπάθειες. Εάν ε, ένα κράτος μέλος ε, δεν πάρει το, από το παράδειγμα μιας ε, μικρής οργάνωσης, έστω μιας μικρής εταιρείας που έχει λειτουργικές δαπάνες κάτω από 7%, τότε ναι να το συζητήσουμε. Αλλά μέχρι τώρα καμία χώρα μέλος δεν έχει δώσει, δεν έχει βρει ένα τέτοιο παράδειγμα. Επίσης, ο μηχανισμός για τη δίκαιη μετάβαση. Ε, παράλληλα έχει ένα ταμείο το οποίο δεν μπορεί να αντιτίθεται στην συνοχή, ένα ταμείο το οποίο δεν μπορεί να αντιτίθεται στις χώρες της συνοχής σε έναν τρόπο κατανομής που επίσης δεν θα πρέπει να αντιτίθεται στις χώρες συνοχής. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά και την ίδια τη σοβαρότητα με την οποία να ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Το InvestEU και η Κεντρική Τράπεζα ε, θα κάνουν μια κατανομή και η ΕΤΕΠ θα πρέπει να κάνουν μια κατανομή σωστή. Ε, δεν υπάρχει earmarking στο InvestEU, δεν υπάρχει earmarking στην ΕΤΕΠ και η ίδια η Κομισιόν έχει κάνει μία, έναν υπολογισμό ε, ανακράτος όμως, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρό. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε στα κράτη-μέλη, δηλαδή ότι θα έχουν ένα τέτοιο ποσοστό ε, ε, και ε, στο οποίο εκεί θα προσθέσουν και ένα άλλο ποσό το οποίο θα προκύψει από τα ίδια τα projects, ένα, ε, θα είναι market driven. Ανώ, είναι ανώφελο να πούμε ορίστε αυτά τα χρήματα θα έχετε γιατί δεν ισχύει αυτό. Είναι κάτι το οποίο στην ουσία οδηγεί σε ανταγωνισμό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και στην ουσία Εάν πούμε το αντίθετο, σημαίνει ότι θα ξαναλλάξουμε την νομική βάση του InvestEU, ενώ εσείς είπατε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η βάση. Και αν δεν αλλάξει η νομική βάση, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κατανομή του InvestEU ε, ανακράτος μέλος, θα μου πείτε βέβαια, είναι απλός υπολογισμός και εκεί μπορώ να συμφωνήσω. Αλλά τότε και εγώ θα σας πω με ποιο τρόπο καταλήγεται σε, αυτόν τον υπολογισμό και ποια είναι ε, τα project που θα πρέπει να υποβάλουν τα κράτη-μέλη. Πράγμα που δεν μπορείτε να μου πείτε, είναι αδύνατο να το ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ευχαριστώ τον Επίτροπο για τη δέσμευση που έχει αναλάβει και εκφράσει. Είμαι βέβαιος ότι θα δουλέψουμε ε, για έναν προϋπολογισμό ε, που έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, είναι ε, ισχυρής θέσης ε, και άλλωστε αποτελεί και την σωστή μεθοδολογία γιατί σε αυτήν την πράξη χρειαζόμαστε όχι μόνο αριθμητικά στοιχεία αλλά και άλλα επιπλέον στοιχεία, το αποτέλεσμα των πολιτικών που επιθυμούμε να έχουμε. Το 1,3 δεν είναι φιλόδοξο. 1,3 είναι αυτό που ζητούν οι πολίτες. Και για να πάω παραπέρα, είναι αυτό που η Κομισιόν ζητάει και αυτό που τα κράτη-μέλη τουλάχιστον στις αρχικές δηλώσεις τους ζητούν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Χάνη, για πέντε δεύτερα. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο δεν ακούνε οι διερμηνείς. Ωραία. Νομίζω ότι αυτή η χορογραφία που είχα αναγγείλει πριν θα πρέπει να αλλάξει, γιατί αν μιλάει ο καθένας τόσο πολύ ε, θα έχουμε πρόβλημα. Ο Επίτροπος ε, Χάν προτιμάει να ακούσει περισσότερες ε, ερωτήσεις και μετά να απαντήσει, γιατί διαφορετικά θα σκοντάψουμε στη διαδικασία. Ε, σας θυμίζω πάντως ε, να μην ξεπερνάτε το χρόνο ομιλίας σας. Η κυρία Γκουαρδία Θαμπάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Είναι γεγονός ότι επιθυμούσαμε να έχουμε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Η κατάσταση του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά περνούν ε, οι μήνες και δεν βλέπουμε μεγάλη πρόοδο ε, και στο Συμβούλιο, αλλά μετά και στις δικές μας ε, συζητήσεις, συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και αυτό με προβληματίζει, γιατί αναρωτιέμαι προς τα πού πάνε, πού βρίσκονται οι συζητήσεις στο Συμβούλιο, γιατί αυτά που ακούμε εμείς δεν είναι πολύ, πολύ φιλόδοξα και αισιόδοξα. Με προβληματίζουν οι συζητήσεις για το πι που α, ε, ακόμα έχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία θα έπρεπε να είναι σημεία συναπόφασης και από την πρώτη κομπόξ μέχρι την τελευταία δεν έχουμε ε, κανένα αποτέλεσμα από αυτές ε, τις συμφωνίες, τις συζητήσεις και ούτε έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο κάποιο από τα σημεία τα οποία νομίμωστε και θεμητά θα έπρεπε να συζητάει με το Συμβούλιο. Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Ε, Ε, και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι εάν θέλουμε να έχουμε ε, καλή και λειτουργική ε, διοίκηση δεν μπορεί να μην αντικαθίστανται αυτοί που βγαίνουν στη σύνταξη ή που φεύγουν. Επίσης, έγινε αναφορά σε ένα ποσό μεγάλο, ένα τρεις. Η Κομισιόν λέει ότι θα χρειαστούν ζητούμε τουλάχιστον 2 δις 700 για την ε, ε, ε, για τα επόμενα χρόνια, αλλά μέχρι το 30 θα έχουμε το πολύ 2 δις 300 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, τα νούμερα δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Μας ενδιαφέρει ε, πώς αυτά τα 3-3 ε, η Κομισιόν προτίθεται να τα βγάλει τη στιγμή που ακόμα μιλάμε για projects. Από το 20 περάσαμε στο 25% ωραία, αλλά δεν είναι όλα αυτά τα χρήματα και εν πάση περιπτώσει δεν είναι φρέσκο χρήμα. Μιλάμε επίσης για το InvestEU που ενδεχομένως αυξήσει το ποσοστό αλλά τα χρήματα είναι τα ίδια. Μιλάμε για την ΕΤΕΠ ε, η οποία ναι υπήρχε ήδη και πριν άρα αυτά τα 2 δις 700 εκατομμύρια από πού τα βγάζουμε. Πώς πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία ε, επιπλέον. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρει το Κοινοβούλιο ή γενικώ να βρεθούν κάποιες νέες, ε, κάποια νέα εργαλεία από τα οποία θα έρθουν να φέρουν περισσότερα χρήματα γιατί διαφορετικά ε, το ε, πι δέλτα πι δεν μπορεί να φτάσει και γενικώ δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το ποσό των τριών, των τριών τρεις. Thank you. Madame Κυρία Γέχη, το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που μπορούμε να έχουμε σήμερα, καθώς επίσης και με την ομάδα διαπραγματεύσεων, γιατί φαίνεται πραγματικά το ενδιαφέρον που δείχνεται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τους Ευρωβουλευτές. Ειλικρινά λοιπόν σας ευχαριστώ. Πολλά ερωτήματα από τη δική μου την πλευρά. Πρώτον, όσον αφορά τους ιδίους πόρους αναφερθήκατε στα εισαγωγικά σας λόγια στο ότι περιμένετε πολλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι θεωρείτε ότι το ζήτημα αυτό, καθώς επίσης και άλλα, θα πρέπει να αποτελέσουν ε, από αντικείμενο σημαντικών ε, εις βάθος διαπραγματεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό σας, το ζήτημα αυτό σας το διαβεβαιώ. Μολονότι βέβαια, κατά την άποψή μας, ε, έχουμε μια κάποια πρόοδο από πλευρά Συμβουλίου μπορείτε εσείς να μας πείτε, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα καταλήξει τελικά στο τέλος της πραγματεύσεων το ζήτημα αυτό και από τεχνικής πλευράς. Όσον αφορά το καλάθι των νέων ιδίων πόρων, που είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της όλης διαπραγμάτευσης. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα συνέργειας που μας δίνει ο κοινοτικός προπολογισμός Από τι ανταλλαγέ που είχα εγώ με τα εμπλεκόμενα μέρη, κατέληξε ο συμπέρασμα ότι η συμβολή από τη χρησιμοποίηση των πλαστικών αποβλήτων έχει προχωρήσει αρκετά. Όσον αφορά την ποσόστοση από το ETS έχουμε προχωρήσει αρκετά. Το ίδιο και όσον αφορά την εισφορά από άλλους τομείς, από τεχνικής πλευράς, εσείς ως Επίτροπος, θα αρκεστείτε τελικά σε, σε έναν δύο μόνο νέους ιδιοσπόρους είσαι σε Φοντελάιεν εργάζεται περισσότερο για την επέκταση του ETF. Πώς μπορεί να επηρεάσει τους ιδίους πόρους ο τομέας αυτός. Και όσον αφορά άλλους νέους ιδίους πόρους, θα μπορούσατε να μας προτείνετε κάποιες νέες ιδέες γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι είχατε αναφερθεί σε έναν φόρο μία φορά που θα μπορούσε να προκύψει από την εσωτερική αγορά. Έχετε ανάλογες προτάσεις να μας κάνετε για να εμπλουτιστεί κάπως το καλάθι των ιδίων πόρων. Ξέρετε επίσης ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον πάγωμα των τομεακών διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσατε να μας πείτε αν υπάρχουν συγκεκριμένα κράτη-μέλη τα οποία απευθύνθηκαν σε εσά θεωρώντας ότι η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν σκόπιμη, ζητώντας σας να ασκήσετε σε μας πίεση προκειμένου να αλλάξουμε τη στάση μας. Και κάτι ακόμα, μια πιο γενική ερώτηση αυτή τη φορά. Όταν ανταλλάσσουμε απόψεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με εκπροσώπους της Επιτροπής και των κρατών μελών υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες εκφράζονται από τους μεν και τους δε θα μπορούσατε να μα πείτε εσεί, κύριε Επίτροπε, αν έχετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσείς κάποιε κόκκινε γραμμέ και αν ναι, είναι αυτέ. Ευχαριστώ. Merci, Mr. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Αντρέσεν. Θα μιλήσω γερμανικά. Αξιότιμη Επίτροπε, είχαν ε, και εμείς προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία ε, για το κλίμα. Ε, έχουμε πάει πολύ καθοριστική χρονιά μπροστά μας, το 2020 και σίγουρα ο προπολογισμό και το ΠΔΠ θα παίξουν σημαντικό ρόλο ε, και πρέπει να πετύχουμε την πράσινη συμφωνία. Όλα αυτά σχετίζονται και χρειάζονται προσαρμογές και η Κομισιόν βλέπουμε ότι αντίθετα με πολλά κράτη-μέλη είναι έτοιμη να κάνει τολμηρά βήματα και αυτό μας ικανοποιεί αλλά σίγουρα δεν έχουν ολοκληρωθεί καθόλου μάλιστα οι διαπραγματεύσει για το ΠΔΛΤΑΠΗ. Γι' αυτό όπως και ο συνάδελφος Φερνάντες σας ερωτώ και εγώ ποια είναι η βάση ε, που έχετε ε, για τις επενδύσεις. Ε, Γι' αυτό το 1-3 ε, για την επόμενη δεκαετία που θα χρηματοδοτήσει το Πράσινο Σύμφωνο και τα 7,5 δις ε, για το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Ίδια ερώτηση. Ξέρουμε τι λέει το Ελεκτικό Συνέδριο. 1,2 ε, ετησίως υπολόγιζε το Ελεκτικό Συνέδριο. Πολύ ψηλότερα ποσά. Και είναι διαφορετικά τα στοιχεία αυτά από αυτά της Κομισιόν. Θα με ενδιαφέρει εσείς με ποια βάση αριθμητική δουλεύετε, με ποια ποσά, πώς καταλήξατε σε αυτόν τον υπολογισμό και επίσης ε, το θέμα δεν είναι μόνο τα ποσά, το ύψος των ποσών, αλλά και η ποιότητα. Σας είχα κάνει μια ερώτηση όταν σας πρωτοσυνάντησα στην Ακρόαση πριν από κάποιες εβδομάδες για το climate mainstreaming πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα έργα, τα σχέδια που χρηματοδοτούνται ώστε να είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικά. Άλλοι μιλάνε για τις ε, γεωργικές επιδοτήσεις, έχουμε τα ορυκτά καύσιμα, έχουμε τις ε, υποδομές για τις οποίες πρέπει να γίνουν επενδύσεις και υπάρχει σίγουρα μια ευρεία γκάμα πρωτοβουλειών από πλευράς Κομισιών. Θα με ενδιέφερε όμως μετά την ακρόαση και μέχρι τώρα τι έχει γίνει πάνω σε αυτό αυτό το τομέα, αν έχετε συγκεκριμένες προτάσεις, αν έχετε κάποια πλάνα ε, και πότε θα τα υποβάλλετε. Γιατί νομίζω αυτό σίγουρα ε, θα είναι σημαντικό και για να δεχθούν κάποια κράτη-μέλη στην ε, Ένωση το σχέδιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Να υπάρχουν δηλαδή και κάποια περί... επιχειρήματα που είναι υπέρ της φιλοπεριβαλλοντικής αυτής προσέγγισης. Σας ευχαριστώ, κύριος Κιούς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Χάν. Πραγματικά καλή είναι η δουλειά που έχεις αναλάβει, δηλαδή να τετραγωνίσεις τον κύκλο. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό με αυτές τις νέες προτεραιότητες και ταυτόχρονα περικοπές σε παλές πολιτικές που μπορεί να μην είναι ίσω ε, πια τόσο σημαντικέ. Θα το δούμε αυτό. Δεν ξέρω αν το πετύχει αυτό θα σε, ε, υπο... θα σε προτείνουν υποψήφιο για το Νομπέλ. Τέλο πάντων, λοιπόν, ας πούμε τη οικονομία έτσι, εντάξει, της οικονομίας. Λοιπόν, νομίζω ότι σίγουρα οι περικοπές δεν μπορούν να αποφευχθούν. Ε, γι' αυτό είμαι πεπισμένος. Αν θέλουμε, μάλλον αν δεν ε, πάρουμε νοπό χρήμα, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες προς αυτό, αυτοί οι οποίοι δίνουν χρήματα αντιδρούν ε, και έχουν επιφυλάξεις. Πώς θα τους πείσουμε ότι θέλουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Και αν δεν τους πείσουμε, σίγουρα οι περικοπές είναι ένα αναγκαίο κακό. Σίγουρα ε, ζητήσατε και εσείς την βοήθειά μας, αλλά ε, δεν μπορούμε να πιστέψουμε και να ορεινερευόμαστε ότι μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι επιτυχίες σε ένα τόσο τεράστιο πεδίο ε, όσο είναι αυτό της οικονομίας, της συνοχής. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα χωρίς περικοπές και Νομίζω ότι και στη ε, διοίκηση πρέπει να υπάρξουν οικονομίες. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο, νομίζω θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε περικοπές. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ελπίζω να μπορέσετε να ε, έχετε αίσιο σε όλες αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις και πραγματικά θέλουμε να ακολουθήσετε μα διαρθρωμένη, δομημένη προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις για να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα δεν θα είναι όλοι ικανοποιημένοι 100% στο τέλος, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια αποδεκτή συνολικά λύση. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ζόνσκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα πολωνικά. Κύριε Επίτροπε, πολύ χάρηκα ε, όταν σας άκουσα στην ακρόαση πριν γίνετε επίτροπος μας είχατε πει τότε ότι θα προσπαθήσετε να προστατέψετε και τις, το Ταμείο Συνοχής ε, και την, ε, τους σιδηροδρόμους ε, προερχόμενους και από την περιοχή των Καρπαθίων. Μπορώ να σας πω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα και εκεί έτσι ώστε να προστατευτεί η περιοχή των Καρπαθίων και σας ευχαριστούμε για την, για τη νέα πράσινη συμφωνία που πολλά μπορεί να προσφέρει σε εκείνη την περιφέρεια. Ρωτώ, θα υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασεων και δράσεων στην περιοχή των Καρπαθιών, ε, ας πούμε έτσι ώστε να αναπτυχθούν ε, ε, διάφορες περιφέρειες εκεί ε, οι οποίες ε, χρήζουν ε, οπωσδήποτε βελτίωση των διαστηνοριακών υποδομών. Επίσης και η χώρα σας και η δικιά μου και καμιά δεκαριά άλλες χώρες λειτουργούν στο τομέα των τριών ε, ευρωπαϊκών θαλασσών ε, και ε, βλέπετε κάποια δυνατότητα υποστήριξης αυτών των σχεδίων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδημού. Mr. Han, please use your headphones until you could learn Greek. Θα τα πω στα ελληνικά. Αν δεν έχετε μάθει ελληνικά, βάλτε τα ακουστικά σας. Καλώς ορίσατε. Είσαστε παλιό, αλλά με καινούρια καθήκοντα πια ω Επίτροπος προπολογισμού. και το πρώτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι δεν είσαστε απλώς honest broker. Είσαστε η Κομισιόν η οποία κατέθεσε συγκεκριμένους στόχους για τα επόμενα πέντε χρόνια δια της Προέδρου της Κομισιόν στην Ολομέλεια του Κοινοβούλου και για να πάρετε ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπατε θα κάνουμε αυτά και αυτά και αυτά σε πέντε χρόνια. Επομένως, έχετε την υποχρέωση να χρωματοδοτήσετε αυτά για τα οποία πήρατε ψήφο εμπιστοσύνη. Και σας ερωτώ, είναι δυνατόν αυτά που υποσχέθηκε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωκοινοβούλιο η Usher Φόντε Λάιεν να υλοποιηθούν με την πρόταση της Κομισιόν η οποία είναι μικρότερη, χαμηλότερη κατά περίπου 5% από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο αν το αναγάγουμε στο ΑΕΠ των 27 χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς είναι δυνατόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά. Αυτό κατά τα γραφάς το είχε πετύχει μόνο ο Ιησούς Χριστός στο θαύμα στο γάμο εν Κανά. Επομένως πρέπει να μας πείτε πώς θα υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Πώς θα γίνει το Green New Deal. Πώς θα υλοποιηθούν οι πρόσθετες πολιτικές για την ανανέωση χωρίς να την πληρώσει η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική. Σημερίζεστε αυτή τη φράση της μόδας ότι αυτά είναι παλιές πολιτικές όπως μας είπε ο εκπρόσωπος της ακροδεξιάς πολιτικής ομάδας που πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη ή θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις πολιτικές για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή όπως ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επιπλέον πότε θα μας παρουσιάσετε τις προτάσεις της Κομισιόν για νέους ίδιους πόρους. Πόσα, από πού και πότε. Και τέλος, ειδικά για το μηχανισμό δίκτυς μετάβασης, του Just Transition Fund, μπορείτε να μας αποδείξετε ότι αυτά τα 7,5 δις είναι όντως φρέσκο χρήμα. Διότι οι δικοί μου λογαριασμοί λένε ότι κόβεται από την πολιτική της συνοχής πολύ περισσότερα από αυτά που δίνεται στο Just Transition Fund. Ευχαριστώ. Thank We Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα τους συντονιστές που μπορούν να κάνουν σχόλια ή να υποβάλουν ερωτήσεις. Όμως, όμως πριν φτάσουμε σε αυτή τη φάση των ερωτήσεων, ίσω ο κύριος Χάν μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσει και τα σχόλια που άκουσε μέχρι τώρα. Κύριε Χάν, έχετε το λόγο. Ε, ε κοιτάξτε, ε, ο μηχανισμός ε, δικές μετάβασης με το Ταμείο και, το πράσι, και η Πράσινη Συμφωνία είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Η δίκαιη μετάβαση ε, βασίζεται σε τρεις πυλώνες και προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Ο, ο πρώτος πυλώνας είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Είναι κάτι το οποίο δίνει δάνεια ο δεύτερος πυλώνας ε, είναι ε, κάτι το οποίο αφορά και την ΕΤΕΠ, το InvestEU, συγγνώμη, που εγγυάται δηλαδή και παίρνει εγγυήσεις ε, από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και αυτός ακριβώς ο δεύτερος πυλώνας στοχεύει μόνο τα λεγόμενα bankable projects. κυρίως εκεί που μπορεί να παρέμβει η ΕΤΕΠ ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί δηλαδή που χρησιμοποιούνται χρήματα τα οποία ε, έχουν προκύψει από, το, από την μόχλευση του Ταμείου ε, Juncker, όπου μπορεί να συμπεριληφθούν και non-bankable projects. Όλα αυτά βρίσκονται στον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. Ε, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά χρήματα, το πραγματικό φρέσκο χρήμα είναι αυτά τα 7,5 δις. Η ε, Φιλανδική Προεδρία στην τελευταία πρόταση που έκανε αναγνώρισε ήδη το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει, να προκύψει επιπλέον φρέσκο χρήμα. Δεν ξέρουμε πόσο, δεν υπάρχει κάποιο ποσό, αλλά πάντως έχει αναγνωριστεί το γεγονός της ανάγκης ύπαρξης φρέσκου χρήματος. Και βεβαίως το ποσό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά έχουμε ήδη τα 7,5 δις. Και υπάρχει και αυτό το, ο, αυτός ο προβληματισμός σχετικά με τα ε, ποσοστά του Ταμείου Συνοχής και τα ποσά τα οποία ε, θα αφαιρεθούν ενδεχομένως. Ε, κάναμε κάποια επικοινωνιακά, αλλά, επικοινωνιακά λάθη στην αρχή. Πάντως, το γεγονός είναι ότι κάθε χώρα θα έχει ένα συμφωνημένο κατανεμένο ποσό για τα διάφορα διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως για την περιφερειακή ανάπτυξη και για το κοινωνικό ταμείο και το γεγονός ότι προκύπτει ένα ποσό όπου προστίθεται και ο ορισμός αυτών των περιοχών που είναι επιλέξιμες ε, για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και μιλάμε ε, για αυτές ε, οι οποίες έχουν εκπομπές διοξιδίου πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βασισμένη στο NATS, σε νατς 3 και ε, με προσπάθεια να φτάσουμε στο επίπεδο ΝΑΤΣ 2, αλλά πάντως ε, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη εμείς θα μειώσουμε τον αριθμό των περιφερειών ιδεοδός σε επίπεδο ΝΑΤΣ 3, δηλαδή στις πιο μεγάλες περιφέρειες, και ε, κάθε κράτος μέλος έχει κάθε ελευθερία να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία και να τα μοχλεύσει ε, με τα χρήματα τα οποία θα προέρχονται από το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Επομένως, ε, τα υφιστάμενα χρήματα των διαρθρωτικών ταμείων θα δώσουν την δυνατότητα να ε, διεκδικήσει κατά κάποιο τρόπο κανείς το τμήμα του ε, ταμείου, των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, όχι το ανάποδο. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται ε, με μοιρασμένη διαχείριση. Τα κράτη-μέλη, ε, οι περιφέρειες τέλο πάντων, είναι αυτές οι οποίες εν τέλει θα διαχειρίζονται τους πόρους του Ταμείου επί τη βάση ενός κοινού προγράμματος που θα έχει συμφωνηθεί και με την Κομισιόν και που θα διασφαλίζει ότι όντως τα χρήματα επενδύονται ακριβώς για στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Ε, υπάρχουν δύο πεδία παρέμβασης. Ε, τα λιγνητικά, οι λιγνητικές και ανθρακές μονάδες ε, και οι ε, βιομηχανίες ε, οι οποίες είναι εντατικής, εντατικών εκπομπών. Και άρα είτε θα αλλάζει ή το υλικό της παραγωγής ενέργειας, είτε θα μετακυλείται σε άλλες ε, βιομηχανίες. Ε, θα, ε, δηλαδή οι χώρες θα πρέπει να βρουν το σωστό μείγμα ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. Το Κοινωνικό Ταμείο ασχολείται κυρίως με την βελτίωση των δεξιοτήτων. Οι άνθρωποι δηλαδή που χάνουν τη δουλειά τους ενδεχομένως βρίσκουν αποκτούν καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες και μετά με τα άλλα ταμεία βοηθιέται η περιφέρεια η οποία θέλει να τροποποιήσει ε, τις ε, εγκαταστάσεις και τις βιομηχανίες. Με αυτόν τον τρόπο εννοούμε ότι θα ε, μπει καινούριο χρήμα και μετά μπορούμε να κάνουμε και μία άλλη συζήτηση για τον τρίτο πυλώνα που είναι η χρηματοδότηση. Είναι φυσικά, φυσικά ξεκινάμε με κάποιες ε, με κάποιους υπολογισμούς σύμφωνα με διάφορα μοντέλα. Βασιζόμαστε στις εμπειρίες μας. Έχουμε κερδίσει ε, μεγάλη εμπειρία στα πλαίσια του Ταμείου Γιούγκερ σχετικά με την ενδεχόμενη μόχλευση ανάλογα με τις χώρες και τους τομείς. Άρα νομίζω ότι οι υπολογισμοί είναι πολύ σοβαροί ε, και μάλιστα έχουν γίνει μάλλον με συντηρητικό τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι εν τέλει και δεν θέλω και εδώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί όλα θα εξαρτηθούν από ποια χώρα ε, θα επιλέξει, ποιου είδους συγχρηματοδότηση, ποσοστά κτλ. Αλλά ε, εντός του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης ε, θα έχουμε δημιουργία 100 ή 120 δις για τα επόμενα τρία χρόνια και αυτός ο μηχανισμός εντάσσεται ε, στο συνολικότερο σχέδιο της ε, Πράσινης ε, Συμφωνίας. Και εδώ έχουν προκύψει κάποιες παρανομήσεις, γιατί εκεί μιλάμε για ένα, τρεις, για δέκα χρόνια. Έχει προκληθεί κάποια παρανόηση. Ε, εμείς έχουμε υπολογίσει αυτά τα οποία μπορούμε να συνεισφέρουμε από ευρωπαϊκής πλευράς για τα επόμενα 7 χρόνια με το ΠΔΠ επί τη βάση των προτάσεων της Κομισιόν και ακόμα βρισκόμαστε στην, αν όχι στην αρχή τουλάχιστον ε, μεσουσών των διαπραγματεύσεων. Άρα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο φτάνουμε σε αυτό το 1-3 εν τέλει τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζω ε, αφορούν την επόμενη επταετία. Αυτό σημαίνει ότι σε 7 χρόνια μπορούμε να φτάσουμε στα 750 δις επενδύσεων που σχετίζονται με, την πράσινη, με το πράσινο θεματολόγιο. 320 δις Δηλαδή 25% αυτό το κομμάτι ε, της συμβολής του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού στο κλίμα. γιατί το σύνολο είναι περίπου 1.280 βάσει της ε, ε, Κομισιόν. Αν τα μοιράσει κανείς, αν τα διαιρέσει δια 4, το 25% είναι περίπου 320. και έχουμε και περίπου 40 δις ε, για δαπάνες ε, και επομένως ε, συγχρηματοδότηση του κλίματος με περίπου 200 εκατομμύρια και περιβαλλοντικές γενικότερα επενδύσεις της τάξης των 50 δις. Ο μηχανισμός δίκαιης μετάδασης συμμετέχει με 100 δις και 18 εκατομμύρια περίπου από το ETS. Άρα όλα αυτά κάνουν περίπου σαν άθροισμα 750 ε, ε, δις για 7 χρόνια. Και αυτό που κάναμε εμείς, μια και μιλάμε για πολιτικά μηνύματα, είναι ότι ε, στα 10 χρόνια κάνουμε μια αναγωγή για τα για τα υπολοιπόμενα δηλαδή τρία αυτά χρόνια επί τη βάση των όσων θα έχουν γίνει τα πρώτα 7 χρόνια υπό την αίρεση ότι τουλάχιστον οι πολιτικές που θα αφορούν γενικότερα το θέμα της κλιματικής αλλαγής θα συνεχίσουν ακόμα και μετά την εκπνοή της επόμενης δημοσιονομικής περίοδου. Και όπως είπα και προηγουμένως, όλες μας οι παραδοχές είναι συντηρητικές. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε τον υπολογισμό επί τη βάση της δεκαετίας. και επί τη βάση πάντα της ε, ε, εισφοράς ε, το, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αυτά τα τρία-τρεις, όταν μιλάμε για εκατομμύρια, καμιά φορά χάνουμε και τον λογαριασμό. Δεν είναι απόλυτα ουτοπία, γιατί είναι γεγονός ότι έχουμε λάβει πολλές αιτήσει που αφορούν κυρίως τις ε, προτάσεις μας που αφορούν την ταξινομία. Πολλά investment funds, πολλοί επενδυτές ε, πραγματικά θέλουν ε, να μάθουν ποιες ε, είναι οι επενδύσεις, ποια είδη επενδύσεων γίνονται αποδεκτές, ποιες είναι φιλικές προς το περιβάλλον που και αφορούν το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ε, γιατί οι επενδυτές και κυρίως τα επενδυτικά funds θέλουν να αναφέρονται εις την ποιότητα των ενδεχομένων των πιθανών επενδύσεων. γιατί και επενδύσεις για συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλα έχουν όλο και περισσότερες υποχρεώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Επομένως, ναι, μπορεί να είναι υψηλό το ποσό, αλλά παρόλα αυτά αντικατοπτρίζει το ποσό αυτό τις υψηλέ προσδοκίες που έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά πρόσθετε επενδύσει. Αυτό είναι λοιπόν σε γενικές γραμμές όλη αυτή η ιστορία για το επενδυτικό πρόγραμμα ε, της Πράσινης ε, Συμφωνίας. Επίσης, υπολογίστηκε ότι οι επενδύσεις NUL για την ουδετερότητα δηλαδή μπορεί να είναι 200, πρέπει να είναι 260 δις αλλά είναι προφανές επίσης ότι αυτό δεν μπορεί να ε, έρθει μόνο από ενωσιακές πηγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, η χρηματοδότηση δηλαδή θα πρέπει να ειδωθεί ε, σαν μια αρχική επένδυση, χρηματοδότηση η οποία θα κινητροδοτήσει άλλες ε, επενδύσεις. Δεν είναι δυνατόν όλοι, όλοι οι πόροι να πηγάσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμπερίληψή μας όμως είναι απαραίτητη. Όσον αφορά του ίδιους πόρου, αναφέρθηκε και από ορισμένου μεταξύ ημών, ε, ναι, το θέμα των πλαστικών αποβλήτων φαίνεται να ε, βρίσκει μεγάλη συνένεση, όχι όμως ομοφωνία προς ώρας. Πάντως έχει αναπτυχθεί και το ETS επίσης και εδώ υπάρχουν κάποιες νέες ιδέες γιατί και το ETS εξαρτάται αν θα υπάρξει παράταση, αν, θα υπάρξει μάλλον διεύρυνση ε, με τον ε, θαλάσσιο τομέα. Υπάρχουν και άλλες ε, ιδέες για συμπερίληψη και της αεροπλοείας κάποια επιβολή ας πούμε φόρου, επιπλέον φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια, κυρίως για τις μικρές αποστάσεις, έτσι ώστε ε, οι ταξιδιώτες να επιλέγουν περισσότερο το τρένο και όχι το αεροπλάνο. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει προκύψει κάποια συγκεκριμένη πρόταση ιδεοδός. Ε, η πολιτική συμφωνία για το επόμενο πιδελταπή θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία σαφή νομική δέσμευση σχετικά με, τις, ε, με τους ίδιους πόρους για το επόμενο π. Ίσως να μην έχουμε την δυνατότητα να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς ποιου είδους θα είναι οι ίδιοι πόροι, αλλά η ιδεοδόση και αυτό είναι νομίζω ο κοινό μας στόχος και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου, θα πρέπει στο τελικό νομικό κείμενο να, περιλαμβάνει, να περιλαμβάνεται κάτι τέτοιο. Άλλωστε και εσείς ε, είχατε να επικρίνετε την έλλειψη μιας ε, νομικής, ε, νομικά δεσμευτικής πολιτικής συμφωνίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια νομική βάση για κάθε ίδιο πόρο. Επίσης, υποβάλλατε ερώτηση σχετικά με, το, με τις κόκκινες γραμμές μας. Κατά τη δική μου άποψη, νομίζω ότι μετακινούνται οι κόκκινες γραμμές με τρόπον ώστε εάν δεν υπάρξουν αρκετά ε, χρήματα να μην ε, υπάρξει χρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Εάν δεν υπάρχει χρήμα δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε οτιδήποτε και ενδεχομένως ε, θα ε, υπάρξει και κάποια κόκκινη γραμμή ε, όπου πραγματικά δεν θα, δεν θα αξίζει και τον κόπο να γίνει κάποια επένδυση γιατί τα χρήματα δεν θα είναι αρκετά. Θα πρέπει να, κατανοήσουν, να το κατανοήσουν αυτό τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν κράτη που ναι θέλουν παραπάνω δραστηριότητες και επενδύσεις αλλά όχι δεν θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Αν δεν έχουμε χρήματα δεν μπορούμε να δαπανίσουμε χρήματα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι επέτης, δεν τριγυρνώ ε, ως επέτης στις διάφορες χώρες. Εγώ λέω ότι ορίστε, αυτά είναι τα ποσά, αυτοί είναι οι λογαριασμοί, μπορούμε να κάνουμε λογαριασμούς και εμείς και εσείς, ε, αλλά είναι ε, προφανής η κατακλίδα ότι εάν δεν υπάρχουν χρήματα... Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καταλάβουν ε, όλοι και να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Στο πρώτο μισό του προηγούμενου χρόνου αποφασίστηκε ε, η διεύρυνση του Frontex με 10.000 υπαλλήλους παραπάνω. Δεν λέω εγώ αν είναι καλό ή κακό, δεν έχει σημασία. Και έξι μήνες μετά ε, έχουμε περικοπή του προϋπολογισμού για αυτή τη συνοριοφυλακή λοιπά κατά 30%. Δεν είναι δυνατόν να προσλάβει κανείς 10.000 ανθρώπους ε, με αυτό το περικομμένο ποσοστό. Εάν όμως ε, πιστεύουν οι περισσότεροι ότι αυτό είναι δυνατό, ε, τι να σας πω, ας προσπαθήσουν να το κάνουν. Είναι, αυτή είναι η πολιτική ε, απόφαση πάντως που ελήφθη. Εγώ γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συζήτηση σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, τι ε, θέλουμε να κάνουμε και μετά να ξεκινήσει η πολιτική συζήτηση η οποία θα φτάσει στην τελική πολιτική απόφαση. Ε, το να πούμε είμαστε έτοιμοι για το 1% και μετά να δούμε τι μπορώ να πάρω, τι μπορώ να, να έχω για 1% δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ σαφέστατα αυτά που είπατε και νομίζω ότι σε σχέση με τους υπολογισμούς στους οποίους αναφερθήκατε θα θέλαμε να έχουμε και περισσότερα στοιχεία για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τους δικούς μας υπολογισμούς μαζί σας. Δέκα ακόμη συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο καθένας σας θα έχει χρόνο αγόρευσης 1,5 λεπτό μόνο. Αν ε, θέλετε βέβαια να έχει χρόνο να σας απαντήσει έπειτα και ο Επίτροπος. Ο κύριος Όλμπριχτ πρώτος παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πάρω το λόγο διότι ο κύριος Φερνάντες με κάλυψε ήδη με τις ερωτήσεις του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μάρκης τότε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα είμαι τόσο σύντομη και γρήγορη όσο ο συνάδελφος. Ε, τέθησαν όντω κάποιε κέρυε ερωτήσει, αλλά θέλω να θέσω και κάποιε επιπρόσθετε ερωτήσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να περιοριστώ στο χρόνο αγόρευση που μου δώσατε. Ωστόσο, θα ήθελα καταρχά να αναφερθώ στο εξή. Είναι σαφέ. Σαφέ ότι συμφωνούμε για τι προτεραιότητε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι συμφωνούν για κάποιε προτεραιότητε. Το θέμα τώρα είναι η διάσταση του προπολογισμού, το μέγεθο του προπολογισμού. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να βρούμε νέου πόρου, δεν φτάνει το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, το GNI. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί στη στάση μα και πραγματιστέ. Πολύ σωστά είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένε ιδέε όσον αφορά του ιδίου πόρου. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Όσον αφορά τι προτάσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια σας. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να έχουμε μία επίσημη αντίδραση από τη δική σας την πλευρά. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 υπέβαλε μια πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Την προηγούμενη τώρα εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια άλλη πρόταση την πρόταση για τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Πώς ερμηνεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρονική αυτή στιγμή ουσιαστικά. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μιλάμε για ένα ενιαίο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι περιλαμβάνεται τελικά η πρόσφατη αυτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τρίτον, την 1η Φεβρουαρίου έχουμε μια συνεδρίαση της ομάδας των φίλων της συνοχής στην Πορτογαλία μετά από πρωτοβουλία του Πορτογάλου Πρωθυπουργού. Γνωρίζω ότι είναι προσκεκλημένοι και οι επίτροποι να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνεδρίαση. Θέτω λοιπόν το ακόλουθο ερώτημα. Ενδεχομένω το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από εμά ποια είναι η σημασία τη πολιτική συνοχή. Ήσασταν ήδη στο παρελθόν επίτροπο για ζητήματα συνοχή. Και έχουμε δει ότι στα δύο τελευταία πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια η πολιτική συνοχής συνέβαλε πολύ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και στην ψηφιακή προσαρμογή. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει την προσέγγιση αυτή, να ευνοήσει την προσέγγιση αυτή υπέρ της πολιτικής συνοχής και εν γέννη στο μέλλον πώς προβλέπει να μετρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δαπάνες που θα γίνουν για την κλιματική αλλαγή και πώς θα καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε τη διάσταση του κλίματος και της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής στις ε, οριζόντιες πολιτικές δημοσιονομικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Λεβαντόφσκι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε έναν έμπειρο Επίτροπο αρμόδιο για όλα αυτά τα δημοσιονομικά ζητήματα πρόκειται για το δεύτερο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Ήδη λοιπόν μία φορά έχουμε ασχοληθεί με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στα πλαίσια της τρέχουσα συνθήκης και βλέπουμε πολύ συχνά ότι οι κανόνες τελικά είναι πολύ καλοί όσον αφορά την ετήσια διαδικασία, όχι όμως αρκετά καλοί για την πολιετή διαδικασία. Ο Χέρμαν Βαν Ρομπέι στο παρελθόν μας είχε πει στις 8 Φεβρουαρίου ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια διακυβερνητική συμφωνία. Το είχαμε κάνει αυτό στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι δυνατό. Εμείς ψηφίσαμε τον Νοέμβριο του 2013, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το 2014-2015 απολέσαμε κάποια προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί. Ποια είναι η δική σα η προσέγγιση όσον αφορά ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να είναι ρεαλιστικό. Δεν νομίζω το βασικό πρόβλημα ποια είναι το Brexit. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι πώς θα καταφέρουμε να ενσωματώσουμε το, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο όσον αφορά αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια. Έχουμε πραγματικά δέσμευση επίσημη των κρατών μελών για το ποσό αυτό. Έχει δεσμευτεί και η δική σας η κυβέρνηση, η δική σας η χώρα. Γιατί μιλάμε για 7,5 δισεκατομμύρια που έρχονται επιπλέον του αρχικού ποσού που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η αρχική πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας. Πάντως, πολύ φοβάμαι ότι το 2021 το έχουμε χάσει σαν έτος χρηματοδότησης. Πρέπει να δούμε αν τουλάχιστον μετά από το αυτό μπορούμε να έχουμε ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη μίλησαν πολλοί συνάδελφοι πριν από μένα. Θα σας ευχαριστήσω κύριε Χάν που είστε εδώ. Δεν θα πω και εγώ ότι πρέπει να κερδίσετε το βραβείο Νόμπελ, ε, ούτε θα αναφερθώ στον Ιησού Χριστό ε, σε σχέση με το εγχείρημα που έχετε αναφέρετε σε πέρας, αλλά ε, να πω ότι η περίπτωση του κράτους δικαίου, για το μηχανισμό δηλαδή για το κράτος δικαίου. Αυτό σε αυτό θέλω να αναφερθώ. Μπορεί να μας διευκολύνει γενικώ. Ε, νομίζω ότι μιλάμε για ένα θεμελιώδη ζήτημα ε, για το κράτος δικαίου στην Ένωση που μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία για την Κομισιόν και για ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι κοντά στους καθαρός συνεισφέροντες. Και νομίζω ότι μπορεί να προωθήσει τη συνεργασία συνεργασία μας. Ο ε, μηχανισμός για το κράτος δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, σε ό,τι αφορά την αποδοχή ε, των πολιτών που θα είναι έτοιμοι να διαθέσουν χρήματα στον νοσιακό προπολογισμό και βέβαια περιμένουν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα δαπανηθούν ε, δυνάμει κανόνων ε, και για την προστασία του κράτους δικαίου. Τι βήματα συγκεκριμένα λοιπόν θα κάνετε ε, για το ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω ότι έχουμε ευκαιρία με το μηχανισμό κράτους δικαίου στο, σε συνάρτηση με το πιδελταπή. Είναι ευκαιρία αυτός ο μηχανισμός. Ευχαριστώ κύριος Μούρεσαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καλώ ήλθατε στην Επιτροπή μου. Κάποιε σύντομε ερωτήσει και από μένα. Προφανώ η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι δύο σημαντικότατα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εμπίπτουν στο δικό σα το χαρτοφυλάκιο. Πολλή δουλειά λοιπόν πρέπει να κάνουμε από κοινού του επόμενου μήνε. Πρώτον, όσον αφορά το μηχανισμό δίκαιη μετάβαση. Είναι σαφέ ότι θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε πολύ γρήγορα τον τρόπο χρηματοδότησή του προκειμένου να στεφτεί με επιτυχία η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να στεφτεί με επιτυχία και όλη διαπραγμάτευση γύρω από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρώτο ερώτημα. Για το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση, όσον αφορά τον πρώτο του πυλώνα, τι είδου μέτρα προτίθεστε εσεί να χρηματοδοτήσετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα έχουμε μία μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική επίπτωση για τα όσα χρηματοδοτούμε και όχι μόνο βραχυπρόθεσμες επιπτώσει. Για τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα πάντα του Ταμείου Δίκαιη μετάβαση, του Μηχανισμού μάλλον Δίκαιης Μετάβασης, ποια μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου οι χώρε αυτέ που χρειάζονται περισσότερο από όλε τι υπόλοιπε τη χρηματοδότηση, που την χάνει να είναι και λιγότερο αναπτυγμένε από οικονομική πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι χώρε αυτέ θα έχουν πρόσβαση στην τόσο αναγκαία για αυτές χρηματοδότηση χρηματοδότηση. Όσον αφορά τώρα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και επιτρέψτε μου να μιλήσω κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ κύριε Επίτροπε, απευθυνθείτε στο Συμβούλιο και πείτε τους να μην θεωρήσουν δεδομένη την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το να θεωρήσει το Συμβούλιο θα τραβήξει την όλη διαδικασία μέχρι το τέλο, φέρνοντα προτελεσμένο το Κοινοβούλιο, το οποίο με το μαχαίρι στο λαιμό θα πει ναι ή όχι, αυτό είναι λάθο. Επομένω, σταθείτε στο δικό μα το πλευρό, εξηγήστε στο Συμβούλιο ποια είναι η στάση μα και η φιλοσοφία μα, όπω άλλωστε τα εξήγησε πριν από λίγο ο κύριο Φερνάνδε. Είπατε ότι πολλά μπορούσαμε να κάνουμε στο προηγούμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ναι, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι δεν είναι και περισσότερου πόρου. Το προηγούμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή άρχισε να χρηματοδοτεί προγράμματα μετανάστευση, στέρεψε εντελώ ό,τι χρήματα είχε στο αποθεματικό, στον υποτομέα 3. Κάθε χρόνο χρειάζεται να εξηγούμε εμεί όμω στο Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει κανένα χρηματοδοτικό περιθώριο. Γιατί ήδη από το 2015-2016 έχουμε αρχίσει να χρηματοδοτούμε την μετανάστευση. Και για τον ετήσιο προπολογισμό, σα παρακαλώ πολύ, λάβετε υπόψη τι κατευθύνε γραμμέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πείτε στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ασκήσει πολιτική πίεση ήδη στην αρχή της όλης διαδικασίας για τον ετήσιο προπολογισμό. Γιατί αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι εγκρίνουν κάποιες ασαφείς πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, λένε ότι θέλουν μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και έπειτα προχωρούν σε συνεχείς περικοπές για την έρευνα, την επιστήμη και το καθεξής. Σας παρακαλώ πολύ, ας εγκρίνει πρώτα το Συμβούλιο τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και ας δεσμευτεί ως προς αυτές στο πλαίσιο του πλαισίου διαπραγματεύσεων το δεύτερο ήμιση του χρόνου. Και ας μην α, ανοίξει τα χαρτιά του Συμβούλιο τελευταία μόνο στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούσολάγκερ έχει το λόγο. Έχω δύο ε, τομείς που θέλω να καλύψω. Ε, το πρώτο είναι η προοπτική, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο Νομίζω ότι ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, μεταξύ Κοινοβουλίου και συμφωνώ σε κάποιες προτάσεις, αλλά μετά υπάρχουν ε, κάποια διέξοδα. Πώς μπορούμε όμως να τα διευθετήσουμε αυτά τα ζητήματα και πώς μπορείτε να πείσετε για το σύστημα ιδίων πόρων για να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Το δεύτερο θέμα, νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για τη βελτίωση της διαδικασίας. Συμφωνώ και εγώ ότι δεν χρειάζεται κανείς να βραβευτεί με το βραβείο Νόμπελ Νόμπελ να γίνει Ιησούς Χριστός για να ανταλύσει αυτά τα προβλήματα, πρέπει να βρίσκονται και πιο απλές λύσεις φαντάζομαι ε, και ένα από αυτά είναι αυτό το climate mainstreaming. Δηλαδή ήδη σήμερα ε, με τον προϋπολογισμό. Ε, Δαπανώνται κονδύλια, αλλά με λάθος τρόπο. Άρα ήδη μπορούμε να βελτιώσουμε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ήμουν ε, πριν από τα Χριστούγεννα στα ελληνικά νησιά και τα συζητήσαμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θέλουμε εκεί διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διάθεση κονδυλίων για τη μετανάστευση, για το άσυλο, για τον έλεγχο στα σύνορα. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν 7-8 διαφορετικές πηγές χρηματοδότηση, διαφορετικοί κορβανάδε και θα πρέπει ε, να δούμε ακριβώς πώς ε, όλα αυτά ε, υπολογίζονται. Εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες αντίξωες συνθήκες και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Γέσερ. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, αγαπητέ Επίτροπε. Εγώ είμαι εισηγήτρια για το gender budgeting. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο γυναικών και εντό κοινοβουλίου και εκτό που ενδιαφέρονται πολύ για αυτά τα θέματα. Ε, σίγουρα υπάρχει αυτή η δυσάρεστη εμπειρία ε, που έχει κανεί. Ε, να θεωρεί κανείς, ε, παραδείγματο χάρη, ότι υπάρχει αρμοδιότητα ε, στι προπολογισμού και μου λένε όχι πρέπει να πάτε στη γάμα δέλτα just. Ότι ναι, εμεί ασχολούμαστε, τα μας λένε με τα θέματα τη δίκαιη μεταχείριση, αλλά πρέπει να δείτε με του προπολογισμού τι γίνεται. Πώ θα κάνουμε λοιπόν αυτή την, το gender budgeting με αποτελεσματικότητα. Έχω πολύ απλέ ερωτήσει και πάλι δεν χρειάζεται να είστε ο Ιησούς Χριστός, νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. και θα πρέπει πιστεύω να φροντίσετε να έχει εξειδικευμένο προσωπικό η γάμα δελτα για το gender budgeting. Θα το κάνετε αυτό και δεύτερο. Αυτά τα άτομα, αυτό το προσωπικό θα μπορούσαν να έρθουν εδώ στο Κοινοβούλιο να μας ενημερώσουν για το πρόγραμμά τους και για τα προσώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρμό η προστασία των, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βεβαίως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, και άλλωστε έχουμε θεσπίσει και την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γι' αυτό. Υπό την ηγεσία της κυρίας Κοβέση, το τμήμα καταπολέμησης της απάτης έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 δις ε, για ε, ε, μία αξία περίπου 40 εκατομμυρίων ανά έτος. Ε, η επένδυση ε, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν μάλλον θα έχει θετική επιστροφή για τον προϋπολογισμό. Αλλά φαίνεται ότι ο προϋπολογισμός ή ε, προϋπολογισμοί των προηγουμένων ετών για το 20 και 21 από την Κομισιόν και για το ΠΔΠ δεν εκτιμούν σωστά την αξία της εισαγγελίας. Από τον ε, ε, Νοέμβριο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μέσα σε 10 μέρες 2.000 υποθέσεις γιατί διαφορετικά θα χαθούν τα χρήματα. Και θα χαθούν πολλά χρήματα, λοιπόν, 2.000 υποθέσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 10 μέρες περίπου, για να αποφασίσουν αν θα ξεκινήσει η δίωξη αυτών των ε, ε, υποθέσεων. Δι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον Επίτροπο να δει ε, από κοντά τις πραγματικές ανάγκες ε, και να δει ποια είναι, ποιοι είναι οι πόροι που χρειάζονται έτσι ώστε να καλύψουν σωστά τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ η κυρία Κέλλερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Μηχανισμός ε, ε, συμπερίληψης ε, διοξιδίου του άνθρακος στα σύνορα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος επιτρέπει επιπλέον πόρους αλλά, ζητά, ε, αλλά πρέπει να είναι ενάρετος κατά κάποιο τρόπο από την ίδια την αρχή του. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν διάσταση τιμών, διαφορά τιμών που αφορά ακριβώς και αντιπροσωπεύει ε, την επιβάρυνση λόγω των κανόνων ε, για το ανθρακικό αποτύπωμα που επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει διαφορετικά αυτή η δυνατότητα της μετακίνησης μέσω δέσμευσης ε, του άνθρακα ε, μπορείτε να μας πείτε τι έχει γίνει πάνω στο θέμα αυτό το οποίο είναι επική, δύσκολο ε, και το οποίο μέχρι τώρα μάλλον έχερε συνενέσεως που έχει προχωρήσει σαν ιδέα αλλά όσον αφορά την επιβολή του, την υλοποίησή του χρειάζεται κάποια τεχνολογική εξέλιξη ενδεχομένως ή κάποιες τεχνολογικές δεσμεύσεις γιατί και αυτό ε, ε, εμπλέκεται στον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σταφανότο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες πολιτικές. Ε, μπορεί να υπάρχουν μικρές αλλά πολύ σημαντικές πολιτικές. Το UCPM δηλαδή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικός από 380 εκατομμύρια ε, έχει φτάσει στα 1,4 ε, δις ε, για, το, για την ίδια περίοδο στο νέο ΠΔΠ. Αλλά έστω και αν αυτός ο προϋπολογισμός ο σημαντικός, ε, οι διαδικασίες ε, διαγωνισμών δεν έχουν προχωρήσει. Ε, το 18, τη διάρκεια 18-19 που είναι πάρα πολύ χρήματα που είναι πολύ σημαντικά για την επισκευή των ελικοπτέρων, για την πρόθεση των φαρμάκων, για τις επιχειρήσεις κτλ. δεν έχουν γίνει και θα ήθελα στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο να προχωρήσουν αυτά γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε μια καταστροφή τύπου Αυστραλίας στην δικιά μας περιφέρεια. Αυτό ε, ε, ξέρετε ότι στην Αυστραλία έχουν καεί ε, πολλά εκτάρια που αντιπροσωπεύουν περίπου την επιφάνεια της Αυστρίας και επομένως δεν το θέλουμε αυτό. Ήδη ε, πάρα πολλές ζωές έχουν ε, χαθεί ε, από τις πυρκαγιές. Δεν θέλουμε σίγουρα κάτι τέτοιο. Επομένως, ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε την Κομισιόν ε, να ε, υλοποιήσει την εντολή της, να καλύψει την εντολή της, έτσι ώστε και τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και τα ιατρικά, όλα αυτά που προβλέπονται στην πολιτική προστασία, να προχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον Επίτροπο Χάν, θα ήθελα και εγώ ο ίδιος να προσθέσω κάτι. υπευλήθη το ερώτημα στον πρώτο γύρο κύριε Χάνα, αλλά δεν απαντήθηκε. Αναφερθήκατε... Αναφερθήκατε, λέω, στο InvestEU και στον ε, προϋπολογισμό του. που υπολογίζεται επί τη βάση ε, πόρων ανά ε, κράτος μέλος. Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο ακούστηκε περίεργο και σε μένα και σε άλλους από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί αν θυμάμαι ε, καλά το EU είναι market-based. Επομένως, ε, τι γίνεται εδώ, πώς πηγαίνουμε από το ένα σκέλος στο άλλο. Μήπως μπορείτε να μας τα εξηγήσετε λίγο αυτά και να απαντήσετε και στα άλλα ερωτήματα βεβαίως. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν να αρχίσω απαντώντας την τελευταία αυτή ερώτηση που θέσατε. Στον πρώτο πυλώνα όντως έχουμε κάποια ποσά τα οποία έχουν προδεσμευτεί, ενώ στον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Και δεχομένω να παρέλειψα να το εξηγήσω αυτό στην πρώτη μου παρέμβαση. Αυτό το οποίο θα κάνουμε ιδίως για να βοηθήσουμε τις περιφέρειες εκείνες οι οποίες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, είναι να τις συνδράμουμε και να τις βοηθήσουμε στο να δημιουργήσουν τα απαραίτητα έργα. Αναφερόμαστε λοιπόν σε περιφέρειες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αυτού του είδους την χρηματοδοτική συνδρομή. Ανάμεσα λοιπόν στις περιφέρειες θα υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού και πρέπει να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Προκειμένου όμως να μην επαναλάβουμε, αν όχι τα λάθη, αλλά τουλάχιστον την ε, αρνητικές εμπειρίες μπορεί να είχαμε με το Ταμείο Γιούγκερ, αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη φορά είναι ότι θέλουμε να έχουμε τέτοιες δομές που να μπορούν τελικά να βοηθήσουν τις περιφέρειες και τις αρμόδιες τοπικές αρχές να προετοιμάσουν κάποια έργα, κάποιες προτάσεις έργων που έπειτα θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από εμά. Αυτά τουλάχιστον στην αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα προϋποθέτουν έναν κάποιο ανταγωνισμό. Κατά αυτόν τον τρόπο οι περιφέρειε με την μικρότερη εμπειρία θα καταφέρουν ουσιαστικά να μην υπολείπονται σε σχέση με τι άλλε και να μην ζημιώνονται πολύ. Όσον αφορά τώρα το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση, αναφέρθηκε σε αυτό και η κυρία Μάρκε. οτιδήποτε προβλέπεται για το Ταμείο αυτό έρχεται ω επιπλέον χρηματοδότηση. Αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια στα οποία αναφέρθηκα είναι νοπό χρήμα. Είναι επιπλέον κονδύλια. Αυτό α είναι σαφέ. Η δική μας η πρόταση, μα πάντα η δική μας η πρόταση είναι αυτή. Αυτή σας εκθέτω αυτή τη στιγμή. Και για να γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε στο μέσο των διαπραγματεύσεων και έτσι περνάω και στη δική σας την ερώτηση. Προφανώς είμαι ευγνώμων προς τον Σάρλα Μισελ, ο οποίος άρχισε να ασχολείται δυναμικά με το ζήτημα αυτό, είναι ιδιαίτερα προσιλωμένος πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη, συγκάλεσε συνεδρίαση των ΣΕΡΠΑΣ. Στις αρχές Φεβρουαρίου θα έχουμε και την συνεδρίαση στην οποία αναφερθήκατε. Επομένως θα έχουμε ένα νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, ενδεχομένως και ένα, μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Πάντω το Συμβούλιο αρχίζει και συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο θα πρέπει να επισπεύσει τι διαδικασίε. Αναφερθήκατε εσεί στο χρονοδιάγραμμα τη προηγούμενη φορά και ήδη υπολοιπόμασταν τότε και ξέρω ότι λάβαμε τότε μια απόφαση στις 30, μάλλον στις 13 με συγχωρείτε Δεκεμβρίου, προκειμένου να αρχίσει η χρηματοδότηση του νέου προπολογισμού από την 1η Ιανουαρίου. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα του κράτους δικαίου. Σε όλες τις διαπραγματεύσεις μας θίγουμε το ζήτημα αυτό. Θα έλεγα ότι ε, είναι μια απέτηση η οποία προέρχεται και από τους καθαρούς εισφορείς Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι σαφώς υπέρ του κράτους δικαίου, ένθερμοι υπέρμαχοι, άλλες λιγότερο, άλλες επιμένουν περισσότερο στο ζήτημα της συνοχής. Έναν κάποιο συμβιβασμό πρέπει να βρούμε ανάμεσα σε όλες αυτές τις χώρες. Και υπάρχει και ένα στερεότυπο, σύμφωνα με το οποίο οι χώρες οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα ταμεία συνοχής, είναι οι πιο ευάλωτε, αν θέλετε, στο ζήτημα του κράτου δικαίου. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2019 αποφάσισε ότι από το 2020 και μετά θα υπάρχει ένας πίνακας αποτελεσμάτων για το κράτος δικαίου που θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη βάσει ισότιμης μεταχείρισης προκειμένου να καταφέρνουμε να εντοπίζουμε αδυναμίες όπου αυτές εμφανίζονται στον τομέα του κράτους δικαίου. και πολλές χώρες να γνωρίσουν από μόνες τους ότι έχουν αδυναμίες και ενδεχομένω οι αδυναμίες αυτές να εμφανίζονται τελικά λίγο πολύ και σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα είναι απόλυτα σκόπιμο θεωρώ να έχουμε μία ομοιόμορφη προσέγγιση για την προστασία του κράτους δικαίου και κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να έχουμε και μια ειδική διακριτική μεταχείριση υπέρ ορισμένων χωρών. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο ισότιμη αντικειμενική μεταχείριση απέναντι σε όλες τις χώρες όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των δαπανών για την πολιτική μετανάστευση και πώς οι δαπάνες αυτές κατανέμονται από τον έναν υποτομέα στον άλλο στον προπολογισμό. Στην τρέχουσα αυτή περίοδο όντως χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή για πρώτη φορά. Στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο βλέπετε ότι προτείνουμε ένα νέο τομέα όπου λέμε ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένε δαπάνε που θα έχουν να κάνουν με την πολιτική μετανάστευση και τα σχετικά ζητήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο στον προπολογισμό και μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα τι σχετικέ δαπάνε και μπορείτε και εσεί ω Κοινοβούλιο να παρακολουθήσετε καλύτερα την κατάσταση. Όσον αφορά το gender budgeting, ο Γενικό Διευθυντή μόλι τώρα με ενημέρωσε ότι θα αναλυφθεί μια σχετική πρωτοβουλία ως, ε, από τη Γενική Διεύθυνση Budget, άρα δεν υπάρχει πλέον καμία άλλη δικαιολογία για περαιτέρω καθυστέρηση. Πολύ γρήγορα λοιπόν θα υποβάλουμε μια σχετική πρόταση όσον αφορά την ένταξη των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ισότητα των δύο φύλων στον κοινοτικό προπολογισμό. Τώρα, όσον αφορά το γενικότερο ζήτημα της ενσωμάτωσης της διάστασης της κλιματικής αλλαγής. όλοι μας, αλλά και οι επιμέρους Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει ε, να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με το ζήτημα αυτό και πολύ απόλυτοι. Να καταφέρουμε δηλαδή να δούμε τι σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και τι όχι. Τι επηρεάζει την κλιματική αλλαγή και τι όχι. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 20% του προπολογισμού μα δαπανάται στον τομέα του μετριασμού τη κλιματική αλλαγή. Αν όμω πραγματικά θέλουμε να φτάσουμε σε ένα ποσοστό 40% του προπολογισμού τη γεωργία που θα σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, είναι 7% του προπολογισμού του Ταμείου Συνοχή, τότε θα πρέπει να είναι σαφέ και το τι μετράει για την κλιματική αλλαγή και τι όχι. Τι συνεισφέρει και τι δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και απέναντι στα κράτη-μέλη για το ζήτημα αυτό, αλλά περιμένουμε στον τομέα αυτό και μια συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο όσον αφορά τον έλεγχο των επιδόσεων. Να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν όντω κάποιε αδυναμίε σε κάποιου τομεί. Μπορεί να μα βοηθήσει και το ελεκτικό συνέδριο να καταλάβουμε τελικά τι συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και τι όχι. Κυρία Κέλλερ. Εσείς αναφερθήκατε σε έναν φόρο που μπορεί να έχει να κάνει με την ε, συνοριακή μεταφορά εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Απόλυτα λογική πρόταση αυτή θεωρώ και απόλυτα δικαιολογημένη. Είχαμε πει ότι επίσης μια τέτοια ιδέα είναι συμβατή και με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Απλώς πρέπει να εξετάσουμε λίγο περισσότερο το ζήτημα αυτό και ενδεχομένω θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε λίγο περισσότερο τον κανονισμό ETS, του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, ή να βρούμε αν θέλετε κάτι εναλλακτικό το οποίο ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε και να είναι αυτή η εναλλακτική πρόταση, θα πρέπει όντω να αντιστοιχεί στη δική σα την ιδέα να καταφέρουμε να έχουμε επίση ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού και να καταφέρουμε να έχουμε μια ισοστάθμιση ανάμεσα στις χώρες εκείνες οι οποίε είναι πολύ αυστηρέ και προσεκτικέ με τι εκπομπέ του δεξιού του άνθρακα και σε εκείνες οι οποίε δεν έχουν ακόμα συγκεκριμένε πολιτικέ. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία στρέβλωση των τιμών εξαιτία των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, από ό,τι κατάλαβα ε, εσείς και αναφέρομαι στην Ευρωβουλευτή που έθεσε το ερώτημα αυτό, ε, ήδη ε, έχετε έρθει σε επαφή με διάφορες χώρες. Από φέτος ξεκινάει πάντως την ε, λειτουργία του, τη λειτουργία της αρχή αυτή. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, όπως ξέρετε, και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εξ αρχής θα πρέπει να δούμε πόσα άτομα θα χρειαστούμε στα πλαίσια αυτής της αρχής. Χρειαζόμαστε έναν νέο διευθυντή, πρέπει όμως να εντοπίσουμε και τις υπόλοιπες ανάγκες, να δούμε τι απαιτείται και ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα οι συζητήσεις, ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητήσεις που έχουν να κάνουν και με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ε, του Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Όλα αυτά προφανώς θα επηρεάσουν και την τελική απόφαση που θα ληφθεί για τη στελέχωση της αρχής αυτής. Είναι κάπως πρόημο να πούμε αυτή τη στιγμή με απόλυτη σαφήνεια τι απαιτείται και τι όχι. Σαφώς δεν είμαστε κατά πάντως της ιδέας που προτείνατε, το αντίθετο κάνουμε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασκούσαμε πίεση για να καταφέρουμε να θεσπίσουμε αυτή τη νέα εισαγγελική αρχή, η οποία βέβαια θα πρέπει να στελεχωθεί και καταλήλως. Τέλος, όσον αφορά την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Προφανώς θα πρέπει να το εξετάσουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή μια απάντηση. Έχουμε τον μηχανισμό αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και η βασική ιδέα ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν τι δικέ του υποδομέ, τον δικό του τον εξοπλισμό, βάσει τη εθνική εμπειρία που έχει το κάθε κράτο μέλο. Ξέρω για παράδειγμα ότι στι κάτω χώρε έχετε επαρκή εξοπλισμό όσον αφορά την απορρόφηση, αποστράγγιση του νερού, το οποίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα υποφελές για τις χώρες που αντιμετωπίζουν ε, πλημμύρες. Στη δική μου τη χώρα έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία όσον αφορά α, τους, τις κατολιστήσεις, για παράδειγμα. Νομίζω ότι όλες οι χώρες έχουν συσσωρεύσει μια κάποια θετική εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις απαραίτητες υποδομές. Πάντως η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε και παραμένει σε επίπεδο κρατών μελών. Ουδέποτε είχαμε πει ότι θα δημιουργούσαμε μια πανευρωπαϊκή δομή. Η κάθε χώρα, όπως σας είπα, συνεισφέρει βάσει της εμπειρίας που έχει η οποία έχει δημιουργηθεί για την κάλυψη των δικών τη αναγκών. Το σημαντικό να μπορεί η υποδομή αυτή και ο εξοπλισμό αυτό να χρησιμοποιείται σε επίπεδο κράτους μέλους, ενδεχομένω και στι όμορε χώρε σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις σας, για τα σχόλιά σας. Εδώ ολοκληρώνεται το σημείο της μερίσιας διάταξης που προέβλεπε τη συζήτηση με τον Επίτροπο Χάν. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ νέου που ήσασταν εδώ και ελπίζουμε να σας βλέπουμε ως το δυνατόν πιο συχνά ε, όποτε είναι αναγκαίο αυτό. Θα προχωρήσουμε σε δύο λεπτά με την ΕΤΕΠ, που είναι το επόμενο σημείο της διάταξης και όσα μας έμειναν από το πρωί. Uh, Συνεχίζουμε με την ε, ημερήσια διάταξη. Σημείο 14, σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ετήσια έκθεση για το έτος 2019. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κορμό, τον εισηγητή, ε, να μας κάνει μια παρουσία παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, διότι αυτό το οποίο σήμερα με ενδιαφέρει είναι να ακούσω τι έχουν να πούν ε, οι εκπρόσωποι των εφόρων πολιτικών ομάδων ε, και οι ευρωβουλευτές που είναι παρόντες. Είχαμε ήδη μία συνάντηση των σκιωδών. Είχα παρουσιάσει σε αδρές γραμμές ε, το σχέδιο έκθεσης με ένα πρώτο τμήμα για το κλίμα, ένα τμήμα για την εξωτερική δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πτυχή που αφορά τη διαφάνεια και κάτι άλλο που ανησυχεί ορισμένους ε, συναδέλφους, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία. Ποιο είναι ο δικός χάρτης, ε, ουσιαστικά, αν θέλετε, ποια είναι η εντολή για αυτή την έκθεση. Ουσιαστικά, ε, να ακολουθήσουμε τις συστάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνούμε άλλωστε μεταξύ μας, στόχος δηλαδή να ε, γίνει μια κλιματική τράπεζα η ΕΤΕΠ και πώς θα το πετύχουμε αυτό. Είχαμε ακρόαση με τον πρόεδρο τη ΕΤΕΠ την προηγούμενη εβδομάδα, Μα είπε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το κλίμα ε, και να γίνει μια κλιματική τράπεζα και πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και πάνω σε αυτά βασιζόμαστε στην εκθέση μας. Δηλαδή λέμε καταρχάς που βρισκόμαστε και εν συνεχεία αναφέρουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τον μετασχηματισμό αυτό, την αλλαγή σε μια τράπεζα για το κλίμα τη ΕΤΕΠ δηλαδή. Φυσικά θέλω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας, τις κριτικές που έχετε να διατυπώσετε και θα κατατεθούν βέβαια και τροπολογίες που φαντάζομαι ότι θα δημιουργήσει, το γεγονός δηλαδή θα μπορούν να συμμετέχουν στην άλλη με θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, ε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, υπάρχει κάποιος από τους σκιώδεις εισηγητές που θα ήθελε το λόγο να παρέμβει. Okay. Oh, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αλλά θα μιλήσω πορτογαλικά. Εξ ονόματος ε, της Αγγέλικα που είναι η σκιώδηση συγγήτρια για την ε, ομάδα μας. Παίρνω εγώ το λόγο και ήθελα να σας πω ότι σε σχέση με την ΕΤΕΠ πρώτα απ' όλα πρέπει να συγχάρω τον εισηγητή μας, τον κύριο Κορμό. Και από εκεί και πέρα, πώς μπορεί να γίνει πιο πράσινη η τράπεζα, είναι το ερώτημα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και τι ορίζει η συνθήκη ε, δηλαδή ότι πρέπει να προωθήσει, να συμβάλλει την ισορροπημένη ανάπτυξη της ε, στέρικης αγοράς. Και λέει και η έκθεση στο 12 ότι θα πρέπει να απαιτεί από τους ενδιάμεσους πελάτες της ε, να δημοσιοποιούν την έκθεση ορεικτά και θα επιβάλλει περιορισμούς στους ενδιάμεσους λοιπά. Αυτό πρέπει να το δούμε. και υπάρχει και ένα ρίσκο εδώ ότι μπορεί οι ενδιάμεση ε, να αυξηθούν και όλα αυτά ε, θα έχουν σαν αποτέλεσμα η χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ να είναι περιορισμένη. Επίσης, το κλίμα και το κλιματικό, κλιματολογικό πρόβλημα δεν μπορεί ε, να λυθεί μόνο με τη στήριξη της βιομηχανίας. Θα έχουμε μία εκβάθρον αλλαγή αν Πραγματικά υπάρχουν καινοτόμε λύσεις συνολικά στον τομέα της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής και η σταδιακή κατάργηση της χρήσης των ορυκτών ε, καυσίμων ε, θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντα υπόψη το τι συμβάσει υπάρχουν σε ισχύ αυτή τη στιγμή. Είναι θετικό που αναγνωρίζεται η σημασία των ΜΜΕ και ανάγκη πρόσβαση αυτών σε χρηματοδότηση, σε τεχνική υποστήριξη και σίγουρα το νέο ΠΔΠ θα πρέπει να δώσει ε, συγκεκριμένη οικονομική στήριξη στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σίγουρα χρειάζεται και περισσότερο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, διότι νομίζω ότι είναι λίγο πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω αν συγκρίνουμε την Ένωση με τη ΣΥΠΑ. Και το τελευταίο που θέλουμε ο ΕΛΚ να τονίσουμε είναι πως υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που προτείνονται και θα θέλαμε η ΕΤΕΠ να ε, έχει μια πιο ενεργό ε, στάση για την ε, πράσπιση της ενεργικής ασφάλειας και τη στήριξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, η ΕΤΕΠ έχει κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και η Αγγέλικα θα καταθέσει τροπολογίες σε σχέση και με τα σχόλια της παρατηρήσεις της ε, που σας μετέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έροχα είναι Λουόμα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Κορμάου ε, για την ε, πολύ καλή δουλειά που αποτελεί βάση για τη συζήτησή μας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν εγερθεί ε, όπως αφορά κατανομή της, της χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ κλπ. Η εστίαση αφορά θέματα του κλίματος όπως σχετίζονται με το κλίμα και επομένως εμ αυτό εξηγείται και από τα σχέδια της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ίδιας της ΕΤΕΠ όσον αφορά ε, το 50% ε, για το χρηματοδότηση κλιματολογικών θεμάτων. Είμαι σύμφωνος με αυτό και θα πρέπει και η ΕΤΕΠ να δίνει περισσότερες αιτιολογήσεις. Μιλήσουμε πάντω πάντως ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν όπως ας πούμε είναι η συνοχή και η ανταγωνιστικότητα ε, της βιομηχανίας μας. Ε, επίσης, ε, όσον αφορά τις ε, ανισότητες ε, εις ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί και θα πρέπει οπωσδήποτε μέσω της σωστής χρηματοδότησης να απαλληφθεί και κυρίως μέσα στα πλαίσια της δίκαιης μετάβασης και πάντα στα πλαίσια της δίκαιης μετάβασης οι δεξιότητες κλπ. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης, ε, πρέπει να σημειώσουμε ότι η θέση και ο ρόλος της ΕΤΕΠ έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί και στο μέλλον, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αναρωτηθούμε για τα αποτελέσματα ε, αυξημένη ευθύνη θα πρέπει να ακολουθείται και από αυξημένο έλεγχο Επίσης ε, πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ όλων των ε, πολιτικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, πρέπει πάντα να εστιάζουμε στα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς που αποτελούν τομείς χρηματοδότησης δανεισμού της ΕΤΕΠ και να δούμε πού υπάρχουν απώλειες ή αποτυχίες αγοράς κλπ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα μέσα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιδιωκόμενων στόχων μέσω των προγραμμάτων της ε, ΕΤΕΠ. Ε, κυρίως ε, πρέπει να δούμε δε και αυτόν τον, την εντολή εξωτερικών δανειοδοτήσεων. Αυτό κατά την άποψή μου θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Ο κ. Χόγης στην προηγούμενη συνάντηση με τούτη την Επιτροπή ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ένα τομέα που εστιάζει την προσοχή της ε, η ΕΤΕΠ. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συσχετισμός ανάμεσα στη χρηματοδότηση τους εξωτερικούς στόχους πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, θα πρέπει να ενισχυθεί η διακυβέρνηση, η καταπολέμηση απάτης, νομιμοποίησης παρανόμων προσόδων κλπ και προσβλέπω σε μελλοντική συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ εγώ, σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι η έκθεσή του αποτελεί πολύ καλή βάση, λέει ο κύριος Χόζικ αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητηθεί καλύτερα είναι ε, η ε, ε, πολιτική συνοχή σε διασύνδεση με την δανειοδότηση, γιατί η ΕΤΕΠ βοηθάει και στις πολιτικές οι οποίες σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς θα χρηματοδοτηθούν, θα χρηματοδοτηθεί γενικά αυτή η Πράσινη Συμφωνία. Γι' αυτό ε, εγώ επιμένω όσον αφορά την έκδοση πρασίνων ομολόγων. Ε, για να μην πω κιόλα ε, ότι ε, υπάρχει και ένα καλό πλαίσιο στα πλαίσια της ταξινομίας σχετικά με το τι, σημαίνει, τι σημαίνουν οι πράσινες επενδύσεις. Δεύτερον, το θέμα της πολιτικής μεταφορών. Καλό ήταν που ακούσαμε από τον Πρόεδρο ότι προτίθενται να υποβάλουν πρόταση για την πολιτική μεταφορών, αλλά καλό θα ήταν εάν και το Κοινοβούλιο τους πιέσει κατά κάποιο τρόπο ε, να ε, υποβάλουν σε προτάσεις τρίτων σχέση με την κυκλική οικονομία. Ήδη είχαμε το ψήφισμα της προηγούμενης εβδομάδας του Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία που καλεί όχι μονάχα γενικά για κυκλική οικονομία αλλά κυρίως για θέματα μη τοξικών ε, ουσιών. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και προς την Κομισιόν και προς τα κράτη-μέλη ε, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, δηλαδή να είμαστε βέβαιοι να σιγουρευτούμε ότι θα υπάρχουν αρκετά, αρκετοί πόροι και όσον αφορά την προετοιμασία των projects, αλλά και όσον αφορά την υλοποίησή τους. Τέλος, διαφάνεια. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και λατρεύω την ε, ε, σύμβαση Atlas in decision making and access to άρχουσε. Αλλά παρόλε τι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα και στα πλαίσια τη ΕΤΕΠ, πιστεύω ότι πάντα υπάρχει η δυνατότητα βελτίωση. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριος Κιού. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα ε, σήμερα να μιλήσω. Είχα θέσει την προηγούμενη εβδομάδα κάποιες ερωτήσεις ε, ε, και σε ό,τι αφορά αυτές τις νέες ωραίες τιμές που δεν έχουν τεκμηριωθεί από τις επιστημονικές ενδείξεις και γνώμσεις με έχουν λίγο στενοχωρήσει και απογοητεύσει και δεν ξέρω ε, αν θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Ε, το θέμα είναι τι θα γίνει με το ποσοστό αυτό το οποίο θέλουμε ε, να χρηματοδοτήσει το νέο πράσινο σύμφωνο και υπάρχουν αυθαίρετες επιλογές και πραγματικά όλα αυτά μου δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά και δεν ξέρω καθόλου πώς θα δικαιολογήσουμε στην κοινή γνώμη και στους πολίτες αυτές τις επιλογές και αυτά τα νούμερα τα οποία προτείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον εγώ είμαι επόμενο ομιλητή, λέει ο πρόεδρο, ε, Και φυσικά θα πάρω το λόγο. Ε, να πω καταρχά ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κόρμο για τη δουλειά που έχει κάνει ήδη πάνω σε αυτή την έκθεση, που είναι σημαντική και είναι και σχεδόν αυτονόητα αυτά που λέει. Δηλαδή, αν το κλίμα, η κλιματική αλλαγή είναι μείζον στόχο για την Ευρώπη, για την Επιτροπή, τότε είναι προφανέ ότι η ΕΤΕ πρέπει να παίξει το ρόλο τη στο πλαίσιο του τόσο σημαντικού αυτού στόχου. Τώρα βέβαια Έχω να κάνω και τέσσερα σύντομα σχόλια. Το πρώτο είναι ότι θεωρώ πολύ σημαντικό ανεξαρτήτως ε, του πώς ε, θα οριστεί με την ΕΤΕΠ, να κρατήσει το τριπλό α. Ε, αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να παραμείνει τράπεζα, γιατί πέραν του κλίματος θα Υπάρχουν ευτυχώς και άλλα στοιχεία ε, στις πολιτικές και στις δράσεις της ε, τράπεζας, ε, τα οποία θα πρέπει να φέρνει σε πέρας όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προανέφερθηκαν και άλλοι τομείς. Δεύτερη παρατήρηση. Θεωρώ ότι δεδομένου του γεγονότος ότι εργάζεται σε ένα περιβάλλον αγορών η ΕΤΕΠ, δεν θα ήταν σκόπιμο να μπουν περαιτέρω περιβαλλοντικοί στόχοι και οδικοί χάρτες που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο φόρτο ε, στην τράπεζα. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε το γεγονός ε, υπόψη ε, ότι δηλαδή πρέπει να δουλεύει αυτό και υποχρεούται να το κάνει και το κάνει. Δουλεύει σε ένα περιβάλλον αγορών η Τώρα, επειδή είναι κατεπήγον το ζήτημα του κλίματος και της επίτευξης των κλιματικών στόχων, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην επιβαρύνουμε με απαιτήσει υποβολή αναφόρων κατά περίπτωση στην ΕΤΕΠ. Ίσως καλό θα ήταν να γίνει σε πιο ομαδοποιημένο επίπεδο έλεγχος και εξέταση από εμάς εν συνεχεία. Και κάτι ε, άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι φυσικά περιμένουμε να ακούσουμε και τη νέα δανειοδοτική πολιτική της ΕΤΕΠ για τις μεταφορές. Αυτά. Ο κύριος Παπαδημούλης τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Κορμάν και να πω ότι το σχέδιο που μας παρουσίασε είναι μια πολύ καλή βάση για συζήτηση αλλά και για το τελικό αποτέλεσμα που θα πρέπει να επιδιώξουμε. Ε, είμαστε λίγες μέρες μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πριν μερικές μέρες ακούσαμε τον κύριο Χόγερ να μας παρουσιάζει τους στόχους για τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε μια τράπεζα για το κλίμα και νομίζω ότι η έκθεση Κορμάν έρχεται να υποστηρίξει ε, αυτήν την ανάγκη και να την μετατρέψει και σε δεσμευτικούς στόχους. Για να είμαι σύντομος θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζουμε αυτή την καταρχήν απόφαση της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να διπλασιάσει τις επενδύσεις έως το 2025 από το 25% στο 50% για το κλίμα και έχουμε ορισμένες παρατηρήσεις ε, για δύο-τρία πράγματα που νομίζουμε ότι χρειάζεται να βελτιωθούν ή να τονιστούν και θα καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες. Το πρώτο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει, σύμφωνα και με το άρθρο 309, έχει ως καταστατικό σκοπό να ενισχύει και την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. Και εκεί χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερο, με δεδομένες και τις ανισότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνω για παράδειγμα το 2018 οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων κατευθύνθηκαν κατά 57% σε μόλις 6 κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ενισχυθεί η χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕΠ και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η τεχνική βοήθεια και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Το τρίτο είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον τομέα της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Γιατί στο παρελθόν είχαμε και πολλές fake πράσινες επενδύσεις ή αποτυχημένες επιλογές χωρίς να δοθεί μέσω του ελέγχου και η, η σχετική ε, λογοδοσία. Γι' αυτό πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να επιδιώξουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να ενισχύει ε, αυτήν την ε, αναγκαία λογοδοσία. Σε αυτό το πνεύμα θα καταθέσουμε προτάσεις πολύ επικοδομητικά επιδιώκοντας να ενισχύσουμε την έκθεση Κορμάν και όχι να την αποδυναμώσουμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, α ακούσουμε τώρα τον κύριο Γκάμπριελ, ο οποίο είναι εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Κογμό, καθώ επίση και του κοιόδη εισηγητέ που εξέθεσαν τι απόψει του όσον αφορά τι οικονομικέ δραστηριότητε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω ενώπιον τη Επιτροπή σα μετά τον επικοδομητικό διάλογο που είχατε με τον Πρόεδρό μα στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι όντω θίγονται διάφορα κέρια σημεία στη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο, αν μου το επιτρέπετε. Η κλιματική εστίαση τη τράπεζα, καθώ επίση και το πώ μπορεί να λειτουργήσει για την εξωτερική χρηματοδότηση η τράπεζα αυτή. Καταρχά, υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πλήρω και είμαστε πανέτοιμοι να, κάνουμε, να διαδραματίσουμε το δικό μα το ρόλο προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία. Οι νέοι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σα έχουν ε, σταλεί θα πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο το οποίο χρηματοδοτούμε κατά 50% για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2055 και επίσης να καταφέρουμε να συμμορφωθούμε με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων μέχρι τα τέλος του 2020. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο μετασχισμός που απαιτείται προκειμένου να εφαρμόσουμε την Συμφωνία των Παρισίων θα πειράσει κάποιου τομεί περισσότερο από ότι κάποιου άλλου. Γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια του Μηχανισμού Δίκαιη Μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεσμεύεται να αυξήσει τη χρηματοδότησή τη αλλά το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι θα αυξήσει και την παροχή συμβουλών προς τις πιο ευάλωτες ομάδες και περιοχές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο. Αυτές οι πρόσφατες λοιπόν φιλοδοξίες και οι σχετικές αποφάσεις στέλνουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τον κόσμο και ενισχύουν το βασικό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός ηγέτης, έχει ηγετική θέση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και περνά έπειτα στη δεύτερη παρατήρησή μου. Η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικά ένας παγκόσμιος αγώνας. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα, λειτουργήσει ως Ευρωπαϊκή Κλιματική Τράπεζα και ως πιο σημαντικός χρηματοδοτικός φορέας θα πρέπει να έχει θετική επίπτωση στις τρίτες χώρες, τις οποίες χρηματοδοτεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια ξέρετε ότι έχουμε ενισχύσει Πολλέ και διάφορε χώρες με πολύ μικρό κόστο για τον κοινοτικό προπολογισμό μέσω διαφόρων μηχανισμών όπως για παράδειγμα η εξωτερική αυτή εντολή, η εντολή εξωτερικών δανείων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είχαμε δάνεια τα οποία δόθηκαν σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, πάνω από 120 χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση εποφελήθηκαν, έχουν εποφεληθεί από τα δάνεια αυτά και εξακολουθούν και χρηματοδοτούνται. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας συνεκτικότητα ανάμεσα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο θεσμός μας αυτός είναι μοναδικός, καθότι μέτοχοι της τράπεζάς μας είναι μόνο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον πλήρη ελεγχό της και είμαστε ο μόνος χρηματοπιστωτικός διεθνής οργανισμός που έχει διαρθρωμένο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτός μην το ξεχνάμε αν τώρα θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ηγετική θέση σε στόχους όπως η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να έχουμε μια χρηματοδοτική πτυχή η οποία είναι πολύ σημαντική. Άρα πρέπει να έχουμε και μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι, όπως λέγεται και στην παράγραφο 33 του σχεδίου έκθεσης, χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων στα πλαίσια του, μέσου ICI. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε στην αρχιτεκτονική μετά το 2020 προβεβλημένο το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να μπορούμε να χρηματοδοτούμε ή να μοχλεύουμε δραστηριότητες δανειοδοτικές από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη ω προ αυτό υπάρχει μια κοινή κατανόηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχουμε αποφασίσει και συγκεκριμένου τρόπου με του οποίου θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κοινή αυτή κατανόηση φαίνεται επίση και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, καθώ επίση και στην εντολή διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι θα διέπει και τι διαπραγματεύσει που θα ακολουθήσουν. Σα ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να μιλήσω εδώ σήμερα. Προσβλέπω ω εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσουμε μια έχουμε επικοδομητική συνεργασία με τη δική σα επιτροπή και εν γέννη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε, κύριε Γκάμπριελ. Ο κύριο Κογμό τώρα. Θέλετε να πάρετε τον κύριο Αγμό, μάλλον πρώτα, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ το ζήτημα αυτό. Έχω ασχοληθεί πολύ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο παρελθόν ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρόταση γνωμοδότηση, την πρόταση έκθεση μάλλον. Πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ισότιμη δανειοδοτική κατανομή. Δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται τόσα πολλά δάνεια σε έξι μονοχώρε όπω ακούσαμε. Στι αρχέ του μήνα, σε μια συνεδρίαση που έγινε στο Λουξεμβούργο, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και δεν έχουμε την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Αυτό υπόθηκε, αλλά δεν ισχύει αυτό. Ο πρόεδρος Γουαγέ μου είπε ότι ακόμα και στη Γερμανία αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες δεν υλοποιούνται κάποια έργα όπως για παράδειγμα στον τομέα των σιδηροδρόμων γιατί δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Οι εμπειρογνώμονες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που είναι και οικονομολόγοι αλλά και μηχανικοί θέλουν να ασχοληθούν με το πρόβλημα αυτό. Έχουν μια συγκεκριμένη πλέον εντολή οι άνθρωποι αυτοί για την προετοιμασία των έργων. Αυτό φαίνεται και από το σχέδιο της έκθεσης. Θα πρέπει όμως να μπορούμε από τεχνικής πλευράς να μπορούμε να πλησιώσουμε περισσότερο τα έργα αυτά. Να υπάρχει δηλαδή και μια παροχή συμβουλών τεχνικής συνδρομής πέρα από την χρηματοδοτική συνδρομή. Ξέρετε, ο Ρούσβελτ με το New Deal δημιούργησε και μια ομοσπονδιακή υπηρεσία για την υποστήριξη των δημοσίων έργων οι πόλεις, οι περιφέρειες, τα ομόσπονδα, οι ομόσπονδες πολιτείες υπέβαλαν σε κεντρικό επίπεδο τις προτάσεις τους και έπειτα σε κεντρικό επίπεδο υπήρχαν δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές οι οποίοι πλαισίωναν από τεχνικής πλευράς τα προτινόμενα αυτά έργα προκειμένου να ευοδοθούν. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό θα πρέπει να επιτρέψουμε και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει πέρα από την καθαρή δανειοδότηση, να συμβάλλει μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης, τεχνικής, η οποία όμως να σέβεται παράλληλα και το περιβάλλον και στα πλαίσια πάντα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Νομίζω ότι αν δεν γίνει αυτό θα γίνουν πολλές ωραίες ανακοινώσεις σε ευσεβείς πόδι, πόθη χωρίς όμως αυτοί να ευοδοθούν ποτέ. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να εμπνευστούμε από την προσέγγιση ε, New Deal που είχε ο Ρούσβελτ στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ε, ο κύριος Κογμόν, πώς θέλει να πάρει το λόγο για να συνοψίσει. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη στιγμή την συζήτηση, να αντιδράσω, μου το επιτρέπετε, εντάχει στι παρατηρήσει που ακούσαμε. Στους, απευθύνομαι στου κοιόδη συζητητέ, να ευχαριστήσω και την κυρία Αγμό. Όσον αφορά το σημείο 12 της εκθεσής μου και τους φόβους που εξέφρασε ο φίλος κύριος Φερνάντες. Κοιτάξτε, Υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Σε ποιον δανείζουμε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Η βασική ιδέα, και αυτό άλλωστε λέγεται και στο σημείο 12, δεν λέμε στο σημείο αυτό ότι θα πρέπει οι πελάτες να δεσμεύονται για όλε τι δραστηριότητέ τους. Αυτό το οποίο λέγεται στο σημείο αυτό είναι ότι εμείς ως τράπεζα σας βοηθούμε προκειμένου να προβείτε σε μία μετάβαση, προκειμένου να αλλάξετε κάπω τα πράγματα. Άρα πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε κάποιες προσπάθειες, κάποιε μεταρρυθμίσει. Εμεί λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν ερχόμαστε για να επιβάλλουμε κυρώσει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όσοι προτίθεστε να κάνετε προσπάθειε θα ανταμυφθείτε με δανειοδότηση και είμαστε εδώ πέρα για να σα πλησιώσουμε κιόλα από τεχνική πλευρά. Το 12 δεν είναι, αν θέλετε, ένα μέτρο το οποίο θα πέσει σε τσεκούρι και θα αποκλείσει κάποιου υποψήφιου δικαιούχου. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι υπάρχουν κάποιε προποθέσει για να βοηθήσουμε και αυτού που δεν είναι έτοιμου να δεχθούν από εμά δανειοδότηση, συμμορφούμε συμμορφούμενοι σιγά σιγά με τις επιβαλλόμενες από εμάς προϋποθέσεις. Τώρα, όσον αφορά τη διατύπωση, χρησιμοποιήθηκε όντως ο όρος κλιματική τράπεζα. Αλλά επειδή προς τα έξω στα πλαίσια της επικοινωνίας μας θα λέμε κλιματική τράπεζα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι είναι και μία τράπεζα, ένας θεσμός, ο οποίος πλαισιώνει κοινωνικά επίσης κάποια έργα και που ουσιαστικά συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχημένη πολιτική κλιματικής αλλαγής αν αυτή δεν διέπεται από κάποιες αρχές ισοτιμίας. Θα συνεχίσει λοιπόν προφανώ να διαδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσέχοντα όμω όλου ιδιαίτερου ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία, την εκπαίδευση και το κ.ο.κ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταθέσετε τροπολογίε προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε περισσότερο το τμήμα αυτό της έκθεσης. Τώρα όσον αφορά τα δάνεια για τις μεταφορές. Και εδώ πέρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να βοηθήσει να επιτευχθεί ο οικολογικός μετασχηματισμός όσον αφορά τις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο παρελθόν έχει χρηματοδοτήσει μεταφορές τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε κάπως αποφύγει, αν θέλετε. Τις οδικές, για παράδειγμα, μεταφορές, το οδικό δίκτυο γύρω από το Στρασβούργο. Κύριε Κέλλερ, εσεί, γνωρίζετε προφανώς πάρα πολύ καλά την πόλη του Στρασβούργου. Η βασική ιδέα εδώ πέρα είναι να χρηματοδοτήσουμε έργα υποδομών, τα οποία να συνάδουν με το βασικό μας στόχο, την καταπολέμηση δηλαδή της κλιματικής αλλαγή, να έχουμε υποδομές μεταφορών φιλοπεριβαλλοντικές. Τώρα όσον αφορά την κυκλική οικονομία, και όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, το είπε αυτό ο συνάδελφος από την ομάδα Renew και αναφέρθηκε επίσης και στα χημικά προϊόντα. Εδώ πέρα όντως έχουμε ένα κέριο ζήτημα. Μία τράπεζα σαν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να συμβάλλει προκειμένου να αλλάξει το οικονομικό μας μοντέλο και να μην έχουμε τελικά ένα οικονομικό μοντέλο γραμμικό το οποίο να βασίζεται σε μια καθαρά βιομηχανική πολιτική, αλλά ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο να είναι πιο κυκλικό και να λαμβάνει υπόψη και όλα αυτά τα οποία είπατε για τι χημικέ ουσίε. Ξέρω ότι ο Σκιώδη, εισηγητή από το Ρινιού, στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με την πρόταση REACH. Λοιπόν, και τα όσα είχαμε πει τότε θα πρέπει να τα έχουμε τώρα κατά νου όταν μιλάμε για την ε, χρηματοδότηση κάποιων ε, έργων. Άκουσα επίσης και κάποιες παρατηρήσεις από την ομάδα ID για κάποια κριτήρια που ενδεχομένω να παραείνε πολιτικά και το καθεξής. Ε, τι να σας πω τώρα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα πολιτικό εργαλείο. Επομένως, θα πρέπει να αποδεχθούμε το ότι μέσω της δανειοδότησης αυτής θέτουμε και κάποιους πολιτικούς προσανατολισμούς, έναν κάποιον πολιτικό δικό χάρτη. Όσον αφορά την αξιολόγηση τριπλό α, κύριε Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκιο. Όσον αφορά τις συμβατικές κλασικές δραστηριότητες ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, γιατί ουσιαστικά η βαθμολόγηση αυτή αντιστοιχεί και στο κόστος της δανειοδότησης, έτσι δεν είναι και λυπάμαι που η βαθμολόγηση αυτή πολλές φορές εξακολουθεί και είναι πιο σημαντική ή της δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από τη διάσωση του πλανήτη και το καθεξής, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αποδεχθούμε. Ενδεχομένω κάποια στιγμή στο εγγύσει απότερο μέλλον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχοντας μια πιο ενισχυμένη πολιτική, οικονομική ε, επιρροή, ενδεχομένως να μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση αυτή. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να έχουμε φτηνό χρήμα για να το δανείσουμε, προφανώς εξαρτώμεθα και από την καλή βαθμολόγηση. Και μην ξεχνάμε ότι μερικέ φορέ προκύπτει κάτι το παράδοξο στην όλη συζήτηση και νομίζω ότι θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε. Υπάρχει από τη μια αυτό που είπατε εσεί, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να προσέχουμε να μην επιβαρύνουμε από διοικητική πλευρά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με πολλέ υποχρεώσει υποβολή αναφορών, με πάρα πολύ διοικητικό προσωπικό, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ενδεχομένω να μην έχουμε του απαραίτητου πόρου για να χρηματοδοτήσουμε έργα. Προφανώ αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια άλλα βάσιμα επιχειρήματα και νομίζω ότι το είπατε και εσείς και άλλοι συνάδελφοι, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μπορεί να λειτουργήσει πλήρως ως δημοσιονομικό οικονομικό εργαλείο, θα πρέπει να, παρέχει και να έχει μάλλον μια τεχνική πλαισίωση. Άρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να υπάρχει και προσωπικό, το οποίο να μην ελέγχει απλώς που πάνε τα χρήματα, αλλά να μπορεί να αποτιμήσει τελικά πώς λειτουργεί το κάθε ευρώ το οποίο ε, επενδύεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από τεχνικής πλευράς. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός που μπορεί να ξέρει πού αντιστοιχεί το ένα ευρώ το οποίο δίδεται για την δημιουργία ενός δικτύου σιδηροδρομικού. Λοιπόν, είτε θα πούμε ότι είναι καθαρά ένας δανειοδοτικός οργανισμός η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι είναι με ένα οργανισμός που δανειοδοτεί αλλά που παρέχει, που παρέχει επίσης και μία ε, τεχνική πλαισίωση. Και κάτι ακόμα και το λέω προς ε, τον φίλο από την ομάδα των Σοσιαλιστών αλλά και προς τον κύριο Παπαδημούλη είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου το ακόλουθο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επενδύει, να δανειοδοτεί εκεί πέρα που ήδη υπάρχει μια σημαντική δανειοδότηση. Δεν θα πρέπει να έρχεται να επικαλύψει δράσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει μέσω της δράσης της να επενδύει κυρίως σε περιοχές που δεν έχουν δοθεί ακόμα αρκετά δάνεια. Επομένως, συμφωνώ μαζί σας ότι είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα τόσο σημαντικό ποσοστό των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που πηγαίνει σε ένα τόσο περιορισμένο αριθμό κρατών μελών. Νομίζω ότι θα πρέπει μέσω της δανειοδότησης της ΕΤΕΠ να βοηθήσουμε και όλες οι υπόλοιπες χώρες που το έχουν προφανώς ακόμα περισσότερο ανάγκη. Τώρα, ε, ένα ζήτημα επί του οποίου δεν αναφέρθηκα αρκετά Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε και τα οποία δεν έχουμε καλύψει στην έκθεση αυτή οι μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσουν επί του παρόντος είναι τα κράτη-μέλη. Μήπως θα πρέπει στο, μέλος να έχουμε, στο μέλλον να έχουμε και ένα άλλο μέτοχο την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δηλαδή. Μήπως θα πρέπει να διευρύνουμε, αν θέλετε, τη συμμετοχή αυτή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό δεν το έχουμε αγγίξει ακόμα. Έπειτα, τι θα γίνει με την δανειοδοτική επενδυτική που έχουμε στον υπόλοιπο κόσμο, με την, υπόλοιπη αυτή, την άλλη αυτή τράπεζα, της οποίας μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο ρόλος. Πώς θα καταφέρουμε ουσιαστικά να συντονίσουμε ή να διασυνδέσουμε το δικό μας το ρόλο με τις άλλες διεθνείς τράπεζες, οι οποίες δανειοδοτούν σε παγκόσμιο επίπεδο ή διασυνοριακά. Εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο υπόθηκε πριν από λίγο. Πάρα πολλοί μιλάνε για το Green New Deal. Στο παρελθόν όμως το New Deal σήμαινε πολλοί νέοι δημοσιονομικοί κανόνες, πολύ έντονη φορολογία και πολλές νέες επενδύσεις. Αν πραγματικά θέλουμε όμως τώρα, εν έτη 2020, να μιλάμε για, νέο, για ένα νέο deal, θα πρέπει αυτό να πλησιώνεται και από συγκεκριμένε δεσμεύσεις και νομίζω ότι αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε πάντα μια σύγκριση ανάμεσα στο New Deal του Roosevelt και το, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ε, θα πρέπει την ανάλυση να, το πάμε, να την πάμε μέχρι το τέλος βασικά, να καλύψουμε όλες τις δεσμεύσεις σαν αυτές που είχαν αναλυφθεί στα πλαίσια του New Deal. Σας ευχαριστώ πάντως για τις παρατηρήσεις σας και περιμένω τις τροπολογίες σας προκειμένου το κείμενο αυτό να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι ε, για την υποβολή τροπολογιών η προθεσμία λήγει την 28 Ιανουαρίου στις 3 ε, το απόγευμα και ότι η έκθεση θα ψηφιστεί στις 2 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πάμε στην άλλη, σε άλλη περιοχή του κόσμου, στην Κίνα. Και θα συνεχίσουμε την πρωινή συζήτηση Για... Κυρία Κέλλερ, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, γραμματεία, κυρίως τον κύριο Ριπέτς, ε, αλλά και την Γενική Γραμματεία για αυτή την πρόταση επιστολής, η οποία θα περιλαμβάνει τις ε, επιθυμίες της κυρίας εισηγητρίας, καθώς επίσης και της σκιώδους Μόνικα Χολμάγερ, Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιμείνουμε στους προβληματισμούς μας και τα όσα μας απασχολούν, χωρίς όμως να πούμε οτιδήποτε ε, ε, για την ενοικίαση στο Πεκίνο ή Beijing. Νομίζω ότι αυτή μπορεί να είναι μια καλή συμφωνία, εάν συμφωνούν οι συνάδελφοι, δηλαδή οι σκιώδεις συνάδελφοι, ε, νομίζω ότι μπορούμε να προωθήσουμε την πρόταση αυτή και ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε που μας δώσατε αυτό το χρονικό περιθώριο για να το σκεφτούμε. Κυρία Χολμάιερ, θέλετε να το δεχτείτε, θέλετε να πείτε κάτι, να ξεκαθαρίσουμε ότι τώρα θα ψηφίσουμε για το Πεκίνο, για το κτίριο του Πεκίνου και στην επιστολή η οποία αποφασίστηκε, θα αποφασιστεί δηλαδή με την ψηφοφορία, θα αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας. Νομίζω ότι ε, μέχρι τώρα πια θα πρέπει να έχετε λάβει όλη την επιστολή, το επιβεβαιώνετε. Ναι, πολύ ωραία, άρα θα ψηφίσουμε. Όσον αφορά το project του Πεκίνου, ναι, θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είστε όλοι έτοιμοι να ψηφίσετε. Άψογα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και επομένως η πρόταση γίνεται δεκτή, 18 ψήφοι υπέρ, 7 κατά. Α, κάτι δεν πήγε καλά. Πρέπει να προσθέσουμε άλλη μία ψήφο στα υπέρ. Κατάλαβα καλά, κυρία Χολμάγερ, και εσείς θέλετε να ψηφίσετε για την επιστολή. Εν πάση περιπτώσει, ε, σας έχει μοιραστεί την προηγούμενη, το προηγούμενο μισάωρο αυτή η επιστολή με όλα τα σημεία τα οποία είχε αναφέρει η κυρία ε, Χολμάγερ. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν σχετικά με την επιστολή με τον τρόπο με τον οποίο είχαμε συμφωνήσει. Μπράβο και συγχαρητήρια κυρία Κέλλερ. Μη φύγετε. Έχουμε ακόμα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε τα σημεία 10 και 11. Ησυχία παρακαλώ. Σημεία 10 και 11 λέει ο πρόεδρος. Ναι, σημείο 10 για το πρωτοκόλλο συνεργασίας, ε, αλληλευτικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Σενεγάλης. Η κυρία Γουαλμίνη δεν είναι εδώ, άρα κυρία Γουαλμίνη έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πάρω το λόγο εξ ονόματος ε, του εισηγητού κυρίου Πάολο ε, Ντε Κάστρο γιατί ταυτόχρονα λαμβάνει η χώρα η Επιτροπή ε, Γεωργίας και δεν μπορεί να είναι παρόν. Ησυχία λέει ο Πρόεδρος παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν λέει η κυρία Γκάρδια Θαβάλ ότι δεν μπορεί να είναι εδώ ο κύριος Ντεκώστα, γι' αυτό τον αντικαθιστώ. Πολύ γρήγορα γιατί ε, ολοκληρώνουμε τώρα την ε, μια λοιπόν συμφωνία αλληλείας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεγάλης ισχύει από το 2014 απλώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρουσίασε ένα, ένα επιπλέον πρωτόκολλο για πέντε χρόνια όσον αφορά τη αλληλευτικά σκάφη ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η νέα πρόταση βασίζεται σε επιστημονικές ε, ενδείξεις. Έγιναν πάρα πολύ μεγάλη και τεκμήρια. Ε, έγινε πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία μεταξύ των αρχών της Ενεγάλη και Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρωτόκολλο. Μιλάμε για 1,7 ευρώ τον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια καθώς επίσης και 900.000 που θα πληρώσουμε όσον αφορά την σαν αντιπαροχή για την εφαρμογή αυτής της ελληνικής πολιτικής. Θεωρούμε ότι το πρωτόκολλο είναι θετικό και επομένως ο εισηγητής ε, σας προτείνει να το υποστηρίξετε και να το υπογράψετε. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος από τους σκιώδεις θέλουν, ε, θέλει μήπως να πάρει το λόγο. Κυρία Λαπόρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτή την ναυτική Συμφωνία υπάρχει ένα σημείο που με προβληματίζει. Απεδείχθη ότι η ε, εντατική αλληλεία των ε, ευρωπαϊκών σκαφών δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την ε, βιοτεχνική αλληλεία ε, της ε, περιοχής. Ε, μιλάμε για την παραδοσιακή αλληλεία των παραδοσιακών αλληλείων της περιοχής που θα πρέπει να προστατευτούν. Άλλα σχόλια. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι αφού δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, στις 17 Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί η γνωμοδότηση. Επόμενο σημείο είναι το πρωτόκολλο για τις αλλιευτικές ικανότητες και την ε, οικονομική συμβολή στα πλαίσια της αλλιευτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. Κύριε Γκερέρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η υφιστάμενη συμφωνία εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας ξεκίνησε το 2016. Στόχος όμως ε, του πρωτοκόλλου είναι να δοθεί ελευτική ικανότητα ε, στα μαυρετανικά ύδατα ε, λαμβάνοντα υπόψη είναι τις διαθέσιμες επιστημονικές, μάλλον τα επιστημονικά διαθέσιμα τεκμήρια έχουμε και την, ε, άλλωστε την γνωμοδότηση της ε, Διεθνούς Επιτροπής Διατήρησης των Θηνοειδών του Ατλαντικού ε, θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια εταιρική σχέση έτσι ώστε να γίνει βιώσιμη η αλληλεία και να υπάρξει βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων. Το τελευταίο πιο πρόσφατο πρωτόκολλο ε, εξέπνευσε το Νοέμβριο του 19. Αυτό το πρωτόκολλο τροποποιήθηκε δύο φορές. Δεν κατέστη δυνατόν η ανανέωση, κατέστη δυνατή η ανανέωση της ε, ε, εταιρική σχέσης, ενώ η Κομισιόν διαπραγματεύτηκε με την Μαυριτανία μέσω, αποστολή, μέσω ανταλλαγής επιστολών. Διαπραγματεύτηκε, λέω, την παράταση του πρωτοκόλλου για ένα έτος. Ανανεώνεται λοιπόν για κατά μέγιστον ένα έτος. Ε, το πρωτόκολλο 1 εκατομμύριο λοιπόν και 12 μήνες επί τη βάση 2 ε, δύο σημείων 57 εκατομμύρια για, τις για τους αλλιευτικούς πόρους για αυτή είναι την 12μηνη περίοδο ανανέωσης καθώς επίσης και υποστηρίξη της αλληλευτικής δραστηριότητας της Μαυριτανίας. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τα θέματα της ε, βιωσιμότητας των αλληλευτικών ε, ε, πόρων της χώρας για όλη την περίοδο εφαρμογής του πρωτοκόλου. Ε, θα πρέπει η υπογραφή να γίνει πριν από την προτινόμενη παράταση ε, Επομένως, η Επιτροπή Αλίας, που είναι αρμόδια ε, επί της αρχής, ζητά να εγκριθεί αυτή αυτό το πρωτόκολλο ε, με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ Μαυριτανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όπου καθορίζονται και οι αλληλευτικές ικανότητες και η οικονομική αντιπαροχή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης η, Επιτροπή Αλίας θα διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό ε, τρόπο αυτή η παρατηνόμενη συμφωνία ε, και με τρόπο ώστε να επιτραπεί ε, η διατροφική κυριαρχία καθώς επίσης και η επιβίωση των αποθεμάτων. Αυτά. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να πάρει το λόγο κάποιος από τους σκιώδεις ε, εισηγητές ε, Στεφανούτε. Πολύ γρήγορα, Πρόεδρε, για να σας πω ότι συμφωνούμε με τα συμπεράσματα του εισηγητή. Όντως, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συμφωνία σύμπραξη. Να επιστήσω όμω την προσοχή σα σε ένα άρθρο που εμφανίστηκε στην Guardian, την εφημερίδα, πριν από τέσσερα χρόνια και στο οποίο λεγόταν ότι τα επιπλέον αυτά χρήματα που αναφέρονται εδώ πέρα, τα 4.125.000 για την υποστήριξη των ελευτικών κοινοτήτων και τη διακυβέρνηση ελευτική πολιτική, λέγεται σύμφωνα με την Guardian ότι δεν πήγαιναν στου σωστού δικαιούχου. Δεν ξέρω λοιπόν αν όντω έχουμε ισχυρού εταίρου τη κοινωνία των πολιτών και αν όντω τα χρήματα αυτά τα οποία δίνουμε καταλήγουν στα χέρια των αλλιέων και όντω αν συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τη πολιτική αλλία στη χώρα αυτή. Δεν είμαστε εμεί Επιτροπή Ελία, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Παρ' όλα αυτά όμω μιλάμε για χρήματα, έτσι δεν είναι. Και εμεί είμαστε υπεύθυνοι για τα χρήματα. Άρα θα πρέπει οι πόροι αυτοί να καταλήγουν στου σωστού δικαιούχου. Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια αρνητικά άρθρα στον τύπο. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς. Αν όχι, να σας πω εγώ... Κύριε Γκερέρο, συγγνώμη, δεν σας είδα. Μα συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος. Προφανώς θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους ιδιαίτερος η κατανομή των χρημάτων αυτών και σε ποιους καταλήγουν τελικά και θα πρέπει προφανώς να καταλήγουν στις αλλιευτικές ε, κοινότητες. Και ναι, μπορούμε σχετικά με αυτό να εξετάσουμε και κάποιες τροπολογίες. Και νομίζω ότι θα πρέπει και στο πλαίσιο της Επιτροπής Αλίας να μείνουμε πάρα πολύ στην παρακολούθηση της συμφωνίας αυτής της σύμπραξης, προκειμένου να μην υπάρχει κατάχρηση της χρηματοδότησης αυτής. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με τον συνάδελφο. Πρόεδρος, η γραμματεία μου πενθύμησε ότι δεν προβλέπονται τροπολογίες για αυτή τη γνωμοδότηση. Όχι, μιλάω για τις τροπολογίες που θα κατατεθούν στην Επιτροπή Αλίας. Πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση στις 17 Φεβρουαρίου. Ολοκληρώνεται έτσι η σημερινή μας συνεδρίαση όπου χρειάστηκε βέβαια να περάσουμε από το ένα σημείο της της διάταξης στο άλλο χωρίς να ακολουθούμε την προβλεπόμενη εδώ σειρά, αύριο στις 9.30 συνεδράσουμε πάλι με μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια ακρόαση σχετικά με τους ιδίους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής. Ελπίζω να είστε όλοι παρόντες. Εγώ θα απουσιάζω δυστυχώς την πρώτη ώρα της ακρόασης. Θα φροντίσω πάντως να επιστρέψω στο μότρο δυνατό. Σε εύχομαι ένα καλό βράδυ.